Right, uh, good Καλή σας μέρα, καλή χρονιά. Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω και πάλι εδώ. Σήμερα το πρωί καλούμεθα να ψηφίσουμε. Βέβαια πρώτα έχω να κάνω κάποιες ανακοινώσεις, οπότε μέχρι να τελειώσω φαντάζομαι θα έχουν έρθει και οι υπόλοιποι για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Συνεπώς, να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη πρώτα, παρακαλώ. Εντάξει, έχουμε πει το καλή χρονιά, έτσι, το θεωρούμε δεδομένο, ότι όλοι το έχουν πει σε όλους. Τι, δέκα λεπτά θέλουμε γι' αυτό. Πέρασαν. Λοιπόν, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δεν βλέπω αντιρρήσεις, συνεπώς εγκρίνεται. Ανακοινώσεις του, της Πρόεδρου τώρα. Για τους τριμερείς διαλόγους έχουμε για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό 18 Δεκεμβρίου και μετά 2,8 και 9 Ιανουαρίου, αυτή τη βδομάδα δηλαδή ακόμα. Εκεί συζητήσαμε τα γενικά θέματα των υποθέσεων ε, αυτών, εποπτικού μηχανισμού. Εξετάσαμε το κάθε άρθρο χωριστά μέχρι το άρθρο 4 στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και νομίζω ότι προοδεύουμε αρκετά εκεί που χρειάζονται συμβιβασμοί. Θα συνεχίσουμε βέβαια και με άλλον τριμερή διάλογο την επόμενη εβδομάδα, στις 16 του μηνός το απόγευμα δηλαδή και έχουμε προγραμματίσει επίσης και για τις 23, 24 και 28 Ιανουαρίου επίσης συναντήσεις. Βλέπετε ότι προχωράμε γρήγορα. Άλλη ανακοίνωση τώρα. Τις ρυθμιστικές προδιαγραφές για το ENA. Πριν από τα Χριστούγεννα ζήτησα παράταση ενός μηνός για τον έλεγχο. Επειδή βέβαια κατά τη διάρκεια των διακοπών δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε στον έλεγχο αυτό. Και έτσι λοιπόν το ζητήσαμε αλλά δεν έχουμε ακόμα απάντηση. Προτείνω λοιπόν να προγραμματίσουμε και συζήτηση για τις ρυθμιστικές αυτές προδιαγραφές. Είναι κάτι που θα έπρεπε να κάνει η Επιτροπή μας και πρέπει να το κάνει κάθε φορά που έχουμε λίγο χρόνο και πρέπει να τον προβλέπουμε αυτό το χρόνο για να συζητάμε και ενδεχομένως να ψηφίζουμε εφόσον χρειάζεται. Το Φεβρουάριο στο Στρασβούργο να ψηφίσουμε. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας ε, δώσουμε εν καιρό. Είναι καλό να μπορούμε να έχουμε συζητήσεις και με το συγητή και με τους σκιώδεις και με τη γραμματεία και οποιονδήποτε να έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Ας έρθουμε τώρα στην ψηφοφορία. Πρόκειται για τον εξυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων. Είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Πρόκειται για την έκθεση του Άντολη Σάντσεφ Πρεσέδο. Πώ ψηφίζουμε, το έχω ξεχάσει, φαίνεται πέρασα πολύ καλά στι διακοπέ, λέει η Πρόεδρος. Αρχίζουμε από την παράγραφο 1. Για να δω λοιπόν ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. απόχέ. Αποχές. Παράγραφο Παράγραφος 1α νέα. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Οι το... οι υπέρ. Κατά αποχές. Εδώ θα πρέπει να μετρήσουμε καλύτερα για χρησιμοποιήστε τις κάρτες σας παρακαλώ. Να αρχίσει η ψηφοφορία. Είναι ένας παραπάνω από το Άλντε που ψηφίζει και από το ΕΛΚΑ. Ωραία, πέρα στις ψηφοφορίες. 19 υπέρ και 2, 21 υπέρ δηλαδή και 15 κατά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που έχω. Εγκρίνεται συνεπώς. Παράγραφος 1β νέα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 8 παρακαλώ. Θα προσθέσουμε και δύο όπως είπαμε. Καράς και Τεμπάκερ. 21 ψήφι υπέρ, 17 κατά. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. Παράγραφος 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 Ωραία. Μαζί μέχρι και την παράγραφο 17. Θα ψηφίσουμε μαζί υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνονται όλες. Να κάνουμε το ίδιο και για τις αιτιολογικές αναφορές παρακαλώ, να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Ναι, citations, έτσι, ένα έως και ένα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Και οι αιτιολογικές σκέψεις τώρα μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται και αυτές. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να έχουμε τα ποσά για το τροποποιημένο κείμενο παρακαλώ. Να ξέρουμε ακριβώς τα νούμερα. Είπαμε θα προσθέσουμε και δύο ψήφους υπέρ. Τρεις ψήφοι υπέρ συνεπώς, 3 κατά και δύο αποχές. Μπράβο, Αντολίν. Καλημέρα και από μένα. Συνεχίζουμε την ημέρηση διάταξη και καταρχήκα χρόνια πολλά σε όλους και από μένα. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημέρηση διάταξης που είναι η εξέταση της έκθεσης για το κοινό σύστημα φόρου προσθέμενης αξίας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των κουπονιών. Είναι η έκθεση της κυρίας Γκάλ Πέρες, στην οποία δίνω και το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω το σχέδιο εκθεσής μου. Επιτρέψτε μου να σας δώσω και μια σύντομη σύνοψη των ουσιαστικών θεμάτων τα οποία εμπλέκονται και θα σταθώ σε αυτά τα θέματα κυρίως. Πρώτα απ' όλα, να θέσουμε το ερώτημα του γιατί η Κομισιόν έχει διατυπώσει αυτή την πρόταση καταρχήν. Όπως ξέρουμε οι συνάδελφοι, η χρήση των κουπονίων δεν υπόκειται αυτή τη στιγμή σε αξιόπιστους κανόνες σε ό,τι αφορά την καταβολή φόρου προς τη θέμενη αξίας. Η κάθε χώρα έχει αναπτύξει το δικό της σύστημα και αυτό εξαλλού είναι σαφές από την έκθεση της Κομισιόν δεν υπάρχει εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με τη χρήση των κουπονιών. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα για τις επιχειρήσεις και για τις φορολογικές υπηρεσίες. Καταλήγουμε λοιπόν σε μια κατάσταση που ένα κουπόνι ε, μπορεί να εκδίδεται σε μια χώρα και να χρησιμοποιείται για καταβολή φόρου σε άλλο κράτος. Και το ερώτημα είναι ποιο είναι το κομμάτι του φόρου που θα πρέπει να εισπραχθεί από την κάθε χώρα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η χρήση κουπονίων που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Κατά την άποψή μου η πρόταση την οποία έχει προετοιμάσει η Κομισιόν <clears throat> στοχεύει στο να εξασφαλίσει μια ενιαία διαδικασία για τη φορολόγηση των κουπονιών αυτών. Αυτή η νέα ρύθμιση Θέλει φυσικά να εξαλείψει την διπλή φορολόγηση των κουπονιών και να εξασφαλίσει και μια ασφάλεια σε σχέση με τις υποχρεώσεις ε, φορολογίας. Έτσι θα μπορούν οι επιχειρήσεις να έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα και αξιοπιστία και επίσης θα βοηθήσει μια τέτοια νέα διαδικασία να μειωθούν οι περιπτώσεις διαφθοράς και ε, φοροαπάτης. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά τα, στοιχεία ουσίας της πρότασης της Κομισιόν, εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι καταρχήν ο στόχος πρέπει να είναι η αποφυγή της διπλής φορολόγησης και η μείωση των περιπτώσεων ε, διαφθοράς ή φοροδιαφυγής και επομένως προβαίνει η Κομισιόν στην πρόταση αυτή για να υπάρξει μια εναρμόνιση ώστε όλα αυτά τα κουπόνια να μπορούν να την χάνουν μια ομοιόμορφη φορολογική αντιμετώπιση. Και αυτό δεν θα πρέπει να έχει καμία σχέση με το πού εκδίδονται ή το πού θα πρέπει να καταβληθούν τα κουπόνια αυτά. Επίσης, ε, η μεταχείριση δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το αν τα κουπόνια αυτά αντιπροσωπεύουν προϊόντα η παροχή υπηρεσιών. Ο στόχος λοιπόν αυτής της ε, ρύθμισης είναι ακριβώς να υπάρξει και ένας νέος και ενιαίος ορισμός των κουπονίων. Αυτό αναφέρεται στο άρθρο 30α. Και επίσης θα πρέπει να υπάρξει κάποια διάκριση για τα κουπόνια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν άπαξ ή πολλές φορές και επίσης να γίνει σαφές πού οφείλεται η καταβολή του φόρου προστέμενης αξίας. Εγώ νομίζω ότι η ρύθμιση αυτή και η ενοποίηση των κανόνων για τα βάουτσερ θα μπορούσε να διευρυνθεί στο μέλλον και προς άλλες κατευθύνσεις, δηλαδή προς άλλα, ε, άλλες μορφές τέτοιων ε, εργαλείων όπως είναι τα κουπόνια. Νομίζω ότι ο στόχος είναι πράγματι να εξασφαλιστεί και μεγαλύτερη διαφάνεια και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κουπόνια τα οποία δίδονται σε, σε ομάδες, σε αλυσίδες, να έχουν ονομαστικό χαρακτήρα, να έχουν ενιαία και σαφή αξία και Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της αξίας αγοράς αυτών των κουπονίων, θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής διαφοροποίηση. Και φυσικά υπάρχουν διάφορες μορφές κουπονίων, τα οποία δεν φορολογούνται όταν υπάρχει μια ε, μεταφορά τους από ένα κάτω σε ένα άλλο, όταν αλλάζουν χέρι, Μονάχα κατά την εξαργύρωση των κουπονίων γίνεται η φορολόγησή τους. Επομένως, με τον τρόπο αυτό η δια... τυχόν διαφορά τιμή μεταξύ τη αξίας καταβολής και τη ονομαστικής αξία είναι περιορισμένη. Τα, προ... τα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγαθά ή υπηρεσίε θα αντιμετωπίζονται διαφορετικά και θα φορολογούνται, όπως είπαμε, μόνο κατά τη στιγμή της εξαργύρωσης. Έχω καταθέσει μια σειρά από τροπολογίες για τα θέματα αυτά, με στόχο να εξασφαλίσουμε ένα κοινό και ενιαίο νομικό πλαίσιο, ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν ενιαίες διαδικασίες στα κουπόνια, εάν αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό θα, αν δεν συμβεί, θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει στο να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση ατόμων που έχουν κουπόνια από διαφορετικές προελεύσεις, να υπόκειται λοιπόν σε διαφορετικές ρυθμίσεις, ακόμα και όταν πρόκειται για κουπόνια τα οποία εξαγοράζουν τα ίδια αγαθά και τις ίδιες υπηρεσίες. Και πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί αυτή η εναρμόνιση. Αυτός είναι ένας τομέας ο οποίος απαιτεί εναρμόνιση ώστε να εξαλειφθούν και οι αβεβαιότητες και οι ασάφειες για τα θέματα αυτά. Υποστηρίζω λοιπόν απόλυτα το στόχο της Κομισιόν να θεσπιστεί ένα ενιαίο σύστημα, μία ενιαία ρύθμιση για όλες τις μορφές κουπονίων σε όλα τα κράτη-μέλη και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την <clears throat> Κυπριακή Προεδρία για την ε, υποστήριξη που μου έδωσε και τη συνεργασία της και φυσικά είμαι έτοιμη να ακούσω και τις απόψεις όλων των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Φερέιρα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αντικαθιστώ την ε, συνάδελφό μου η οποία δεν μπορούσε να είναι εδώ που είναι σκιώδης συγγήτρια θα διαβάσω λοιπόν το κείμενο το οποίο μου έδωσε για να το μεταφέρω εξ ονοματός της. Να ευχαριστήσω πρώτα τον, την εισηγήτρια για την εργασία την οποία έκανε όσον αφορά το θέμα αυτό. Η πρόταση της Κομισιόν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός όσον αφορά την εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων ε, και των συστημάτων ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα συμβάλλει βεβαίως ε, στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Ε, ε, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κρίση και λαμβάνοντας υπόψη και την πίεση ε, της ε, δημοσιονομικής εξυγίανσης, το θέμα αυτό γίνεται πάρα πολύ σημαντικό. Στην χρήση των κουπουνιών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και σειρά μελετών που εκτιμούν το βάρος το οποίο έχουν στην εμπορική πολιτική ε, σε πολλά ε, δισεκατομμύρια και βεβαίως θα πρέπει να αποφευθεί οποιαδήποτε προσπάθεια αποφυγής ε, φορολόγησης μέσω των κουπονιών. Καλωσορίζουμε την πρόταση της Κομισιόν διότι προσπαθεί να καλύψει ε, και τον νομικό κατακαιρματισμό καθώς επίσης ε, και τις νομικές ελλείψεις οι οποίες μπορεί να παρουσιάζονται στην νομολογία των κρατών μελών. Ε, με τον τρόπο αυτό ε, δεν καλύπτονται τα προβλήματα φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής. Η θέση της εισηγήτριας ε, με βρίσκει σύμφωνη και θεωρώ ότι η εργασία και η συνεργασία μάλλον στις επόμενες εβδομάδες με την εισηγήτρια θα είναι εξαιρετικά επικοδομητική. Παρ' όλα αυτά παραμένουν κάποια ζητήματα προς επίλυση πριν ε, ε, τεθεί σε ισχύ η οδηγία. Ε, η Σκιώδη Συγήτρια πιστεύει ότι θα πρέπει να εισαχθούν νέα στοιχεία. Πρώτον, η πρόταση αυτή δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα παρομοίων με τα κουπόνια θεμάτων, δηλαδή εκτός από τα vouchers και τα κουπόνια, coupons στα αγγλικά. Θα πρέπει επίσης ε, ε, στην οδηγία να αντιμετωπιστούν και αυτού του είδους ε, τα κουπόνια. Επίσης για την καταπολέμηση της φόρο αποφυγής θα πρέπει να αρθούν τα εναπομείναντα προσκόμματα ε, και ε, κατά αυτήν την έννοια θα πρέπει όλοι οι κανόνες του ΦΠΑ ε, να εξομοιωθούν. Επίσης υπάρχουν παραδείγματα υπερβολικού διοικητικού άχθους ε, κυρίως ε, για κουπόνια τα οποία χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές χώρες μέλη. Κατά την άποψη της σχεδούς εισηγητρίας μπορούν να υπάρξουν απλουστευμένες ε, διαδικασίες. Συγκεκριμένοι λοιπόν απλουστευτικοί κανόνες έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν από τη μία οι διάφορες περιπτώσεις αλλά χωρίς από την άλλη να υπάρξει περαιτέρω σύγχυση. Η σκιώδη εισηγήτρια θεωρεί ότι η πρόταση της Κομισιόνα αποτελεί σημαντικό βήμα προς την την ενοποίηση της ενός αγοράς και ε, προς, το, ε, προς τη κατεύθυνση όσον αφορά τη φορολογική πολιτική. Ε, θα πρέπει κατά την άποψή της η εφαρμογή της οδηγίας αυτής να έχει θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σκιώδης εισηγήτρια ελπίζει ότι θα συνεχίσει με την εισηγήτρια την στενή συνεργασία για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, τους τώρα, κύριε Δηλάκερα. Ευχαριστώ τον κύριο Σκυλακάκη, αντικαθιστό, που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Θα σας διαβάσω και θα κάνω και κάποια σχόλια εκ μέρους του. Και εκείνος θα με ευχαριστήσει βέβαια τον συγκητή για την προσπάθεια που έκανε για αυτό το θέμα. Βασικά συμφωνεί με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύει ότι οι τροπολογίες ε, που προτείνονται είναι λογικέ, αλλά υπάρχουν και δύο σημεία στα οποία θα ήθελα να αναφερθεί και είναι τα δύο εξή. Πρώτα απ' όλα πιστεύει ότι για να ξεπεράσουμε τις αρνητικέ συνέπειες από τον κατακαιρματισμό των κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσουμε ότι την ίδια μερομηνία θα αρχίσει να ισχύει η οδηγία σε όλε τις χώρες μέλη. Βέβαια υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν ήδη Μάλλον αν κάποιες χώρες εφαρμόσουν την οδηγία και κάποιες όλες όχι, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται στρέβλωση. Δεύτερον, υπάρχει κάτι πιο γενικό που έχει να κάνει και με πολλές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει να κάνει και με αυτήν. Συζητάμε πώς θα πετύχουμε μια αυθεντική ε, οικονομική ένωση και νομισματική ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι έτσι επηρεάζονται και οι δημοσιονομικές πολιτικές των χωρών. Αυτό διευκολύνει τη συζήτηση περισσότερο εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πει ότι όλες οι προτάσεις αυτές έχουν τις ίδιες φορολογικές επιπτώσεις και δημοσιονομικές σε όλες τις χώρες. Από εκεί και πέρα είμαστε όλοι διατεθειμένοι να συνεργαστούμε για να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα από κοινού. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριο Στεπάκερ τώρα εκ μέρου των πρασίνων. Ε, που πήρε το εκ μέρου των πρασίνων τώρα των συντηρητικών. Δεν βλέπω κανέναν. Όχι, όχι. Ωραία. Και πάλι λοιπόν η συγκήτρια. Τι έχει να πει για να σχολιάσει τις παρατηρήσεις που έκαναν οι συνάδελφοι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις προτάσεις σας και για την επικοδομητική σας κριτική. Συμφωνώ με τους συναδέρφους για το ότι αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι ότι οι κανόνες ΦΑΠ είναι ε, ομοιόμορφοι, ότι δεν αυξάνουν τη γραφειοκρατία, πράγμα που σημαίνει ότι φυσικά και πρέπει να υπάρξει αναρμόνιση. Θέλω τώρα να αντιδράσω και στα σχόλια των συναδέλφων που είπαν ότι πρέπει να υπάρχει συνοχή στην πρότασή μας. Ε, πράγματι, είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι το είδος της πρότασης που βοηθάει την εσωτερική αγορά να σταθεί στα πόδια της ή την καταστρέφει. Η χρήση λοιπόν των κουπονιών και άλλων ε, προπληρωμένων μέσων είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίζεται ομοιόμορφα παντού. πρέπει να δούμε τι είδους vouchers υπάρχουν για ένα σκοπό, για πολλούς σκοπούς. Είναι μέσα πληρωμής και αυτά που χρησιμοποιούνται στην πράξη σήμερα από πολλούς λιανοπολιτές. Άρα πρέπει να δούμε κατά ποιο σύστημα ρυθμίζονται αυτού του είδους οι πρακτικές. Επίσης να δούμε πώς μεταφέρονται στην νομοθεσία οι κανόνες. Τι δυνατότητες νομικές υπάρχουν και ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων. Γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη θα διαπραγματοφθούν. Αυτό που μπορούμε λοιπόν εμείς να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τους ίδιους κανόνες, να έχουν τους ίδιους ορισμούς. Και όσον αφορά τώρα την ε, έκθεση επιπτώσεων, την έρευνα επιπτώσεων, υπήρξε μια τέτοια μελέτη, μια τέτοια αξιολόγηση και ακριβώς γι' αυτό υποβλήθηκε και η τροπολογία στην αρχική πρόταση. Εγώ δηλαδή πρότεινα να υπάρξει μελέτη. Εξού και η τροπολογία μου. Από εκεί και πέρα είμαι στη διάθεσή σας και στη διάθεση των σκιωδών εισηγητών για να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα να σας πω δύο λόγια παρακαλώ. 23 Ιανουαρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και 18 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε. Και μετά τον Απρίλιο θα πάει στην Ολομέλεια το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Αγκάλ. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 23 Ιανουαρίου. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες 18 Φεβρουαρίου και η ψηφοφορία στην Αρμόδια Επιτροπή είναι στις 25 Φεβρουαρίου και στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της ημέρησης διάταξης, η συζήτηση των τροπολογιών για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σε ό,τι αφορά το συντονισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών η ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη για το 2013. Άνευ καθυστερήσεως δίνω το λόγο στην κυρία Φερέιρα η οποία είναι και σχετικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν συμβάλει στο κείμενο και το έχουν βελτιώσει με τις ε, συμβολές τους. <clears throat> Πάνω από 300 τροπολογίες ε, κατατέθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι επειδή θα πρέπει να διεκπαιρεωθεί αυτή η έκθεση σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εγώ χρειάζεται να καταβάλω μια τεράστια προσπάθεια να συγκεντρώσω τις τροπολογίες αυτές και ζήτησα όμως και από τους συναδέλφους να με βοηθήσουν να επιτύχουμε κάποια σύγκληση για τις τροπολογίες αυτές. Πιστεύω ότι αυτή η σύγκληση απόψεων είναι εφικτή γύρω από μερικές βασικές ιδέες και έννοιες. Δεν μπόρεσα βέβαια με συμβαστικές τροπολογίες να καλύψω όλες τις συνεισφορές των συναδέλφων γιατί υπάρχουν σημαντικές αποκλήσεις μεταξύ των διαφόρων θέσεων. Εξακολουθώ όμως να πιστεύω ότι είναι εφικτό να εξασφαλίσουμε μια αρκετά στερεά και ισχυρή συνένεση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απόψεις των πολιτικών ομάδων και όλα αυτά μπορούν να είναι μια βάση για μια συνολική συνένεση. Για μένα υπάρχουν δύο στόχοι που θα πρέπει να εξυπηρετήσει αυτή η έκθεση. Ο πρώτος στόχος <clears throat> είναι να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια της εκπόνησης της ετήσιας επισκόπησης ανάπτυξης. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί μέσα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο υπάρχουν δύο στιγμές που γίνεται ένας απολογισμός και εξετάζουμε τις μελλοντικές προοπτικές και αυτές οι στιγμές αντιμετωπίζονται στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης, το Annual Growth Survey και επίσης το σημείο το χρονικό που δίδονται οι συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Αυτά τα δύο λοιπόν χρονικά ορόσημα θα πρέπει να μας βοηθούν να έχουμε μια καλύτερη ιδέα για την οικονομική εξέλιξη στη ζώνη του ευρώ αλλά και γενικότερα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλέκεται περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, να έχει μια μεγαλύτερη λοιπόν συμβολή στο να παρακολουθεί την εφαρμογή του six pack του εξάπτυχου ή του μελλοντικού δίπτυχου του pack. Αυτή είναι λοιπόν η στρατηγική έποψη που μου φαίνεται κεφαλαίωδης. Δεν πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα θέματα να την χάνουν συζήτησης μόνο έξω από την, ε, τον ενωσιακό χώρο, από τον έλεγχο του Κοινοβουλίου και χωρίς συμβολή του Κοινοβουλίου και επομένως να εκφεύγει από κάθε δημοκρατικό έλεγχο, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός να ενισχυθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και φυσικά και με τη βάση των προηγουμένων αποφάσεων που έχει λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε σε σχέση με το Six Pack είτε με το Two Pack είτε και σε σχέση με την συζήτηση των συστάσεων που απευθύνονται προς τα κάτι μέλη. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος λοιπόν που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να επιτύχουμε. Ο δεύτερος στόχος είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία ώστε να προκύψει μια σοβαρή συζήτηση η οποία δεν χρωματίζεται ιδεολογικά αλλά που μπορεί να μας βοηθήσει να θέσουμε αντιμέτωπη τη θεωρία με την πραγματικότητα και να έχουμε μια στρατηγική διασταυρούμενων ελέγχων, να μπορέσουμε λοιπόν μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουμε μια συζήτηση πλήρη για το αν είναι επιτυχής και υποφελής πολιτικές που ακολουθούνται και σε ποιο βαθμό θα είχε νόημα να τις τροποποιήσουμε ή όχι για να επιτύχουμε τους τεθειμένους στόχους. Ζούμε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονική συγκυρία, μια κρίση που δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ευρώπη, τουλάχιστον από τότε που υπάρχει το ευρώ, και τα αποτελέσματα τα οποία έχουν ε, προκύψει από την εφαρμογή αυτών των πολιτικών θα πρέπει να είναι αντικείμενα ειλικρινού συζήτηση για να μπορέσουμε να έχουμε πάντα στο μυαλό μας με ποιο τρόπο μπορεί να τροποποιηθεί η γραμμή πλεύσης που έχει ακολουθηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα οικονομικά αυτά θέματα. Εγώ θεωρώ ότι από την πρόταση της Κομισιόν έχουμε πέραν της τη Κομισιόν έχουμε και την τεχνική εργασία που προέρχεται από τρεις χώρες που εργάστηκαν από κοινού. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν <clears throat> στον έλεγχό μα, και κατέδειξαν αυτές οι, αυτά τα στοιχεία ότι εφαρμόστηκαν ορισμένε διατάξεις με υπερβολική πίεση και όχι με την απαραίτητη ε, αντιμετώπιση τόνισαν πάρα πολλοί οικονομολόγοι ότι έχει υποτιμηθεί η ο υφεσιακός αντίκτυπος αυτών των μέτρων και επομένως εν μέρει αυτά τα μέτρα είχαν ένα αντιπαραγωγικό χαρακτήρα. Αυτό μας υποχρεώνει να χρησιμοποιήσουμε το περιθώριο ελιγμών που έχει δημιουργηθεί μέσα στο six μέσα στα πλαίσια μιας οικονομικής κρίσης, όταν τα αποτελέσματα των μέτρων που λαμβάνονται έχουν ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά λοιπόν μας οδηγούν στο να κάνουμε αυτή την άσκηση η οποία πρέπει να είναι και μια άσκηση ευθύνης. Μέσα στα πλαίσια αυτά λοιπόν πιστεύω ότι υπάρχουν ορισμένα επιμέρους θέματα τα οποία καλύπτονται σε αυτή την έκθεση. Καταρχήν, μια περιγραφή του πώς προέκυψε η κρίση που είναι σημαντικό γιατί η αντίληψη της, ε, του τρόπου με τον οποίο προέκυψε η κρίση θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς θα τη θεραπεύσουμε. Υπάρχει εδώ ένας μεγάλος αριθμός τροπολογιών για το σημείο αυτό, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε με τους κοιόδης συζητητές να καταλήξουμε και σε κάποια μεγαλύτερη συνένεση στα διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τη περιγραφή του πώς έλαβε χώρα η κρίση και ποια μορφή έλαβε. Επίσης μέσα στο ίδιο αυτό πλαίσιο θέλουμε να βρούμε και κάποια σημεία επαφής, κάποια σημεία συμφωνίας σε σχέση με την ανάλυση των πολιτικών που ακολουθήθηκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης, κάτι το οποίο ενδεχομένως θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε και σε μια μεγαλύτερη συμφωνία, μια μεγαλύτερη συνένεση για το αν οι πολιτικές αυτές είναι απόλυτα ορθές ή αν χρειάζεται να υπάρξει μια τροποποίησή τους ή αν χρειάζεται <clears throat> να παραταθούν ορισμένα από αυτά τα μέτρα για να μπορέσει να υπάρξει μια διόρθωση στα δημόσια οικονομικά των χωρών της ζώνης του ευρώ που να είναι λιγότερο βία και να έχει λιγότερο αντίκτυπο. Επίσης έχουμε θέματα τα οποία συνάπτονται με τις ε, κατεπίγουσες δράσεις οι οποίες χρειάζεται να αναλυφθούν. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να θέσουμε να ανακλήφο κυρίως στο θέμα της ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων, ως ένα από τους τομείς, ως τον τομέα που πρέπει να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατό. Και είναι απαραίτητο να βρούμε μια λογική συνένεση γύρω από το θέμα αυτό με τις διάφορες πολιτικές ομάδες, ε, παραγωγός με τις προτάσεις που έθεσε ο κύριος Κλίντς ή η Πράσινη ή κάποιες από τις προτάσεις του ΕΛΚ. Ο αγώνας επίσης έναντι της ε, φοροδιαφυγής και της φοροαπάτης πρέπει να τύχει αναγνώριση από όλους μας ως ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί είναι κάτι το οποίο μειώνει και την νομιμοποίηση των πολιτικών λιτότητος που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δημιουργείται η αίσθηση στον πληθυσμό ότι υπάρχει μια θεμελιώδης αδικία όταν επιτρέπεται λόγω ανικανότητος ή λόγω ανοχής να μπορούν να διαφεύγουν φορολογήσιμα ποσά <clears throat> και να διαφεύγουν πολλοί πολίτες από τις υποχρεώσεις τους ενώ άλλοι πολίτες βρίσκονται σε κατάσταση ένδυας. Και εδώ έχουν κατατεθεί προτάσεις από τον Έπινγκ, την Βόρτμαν, Κόλ που βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσε, από τον κύριο Μπουλάρ επίση και πιστεύω ότι και εδώ μπορούμε να συγκλίνουμε με κάποιο τρόπο στην ε, περιγραφή αυτού του προβλήματος. Για το δημόσιο χρέος επίση. Μπορούμε να επανέλθουμε και να υπενθυμίσουμε αυτά τα οποία έχει πει η Επιτροπή μας σε προηγούμενα κείμενα. Και επίσης νομίζω ότι μπορούμε να τονίσουμε τον κεντρικό αυτό στόχο του να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα πολύ πιο ενεργό ρόλο από ό,τι είχε μέχρι τώρα για τα θέματα της αξιολόγησης του δημοσίου χρέους και επομένως να έχει μια συμμετοχή και να μπορεί να ασκεί κάποια επιρροή στη διαμόρφωση της ετήσιας επισκόπησης ανάπτυξης και των στρατηγικών που έλκονται από αυτή την έκθεση. Για όλους αυτούς τους λόγους αυτό το οποίο θα προσπαθήσω να κάνω είναι στην αρχή της επόμενης εβδομάδας να μοιραστώ με τους συναδέλφους, να διανύμω καλύτερα στους συναδέλφους μια πρώτη προσπάθεια, ένα πρωτόλιο σχέδιο προσπάθειες εξέβρεσης συμβασμού, γνωρίζοντας ότι το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σφιχτό και πρέπει να υπάρξει και μια ταχεία αντίδραση των συναδέλφων σε αυτό το πρώτο σχέδιο για να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές λύσεις και θεωρώ επομένως ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε μετά στις προσπάθειες να καταλήξουμε σε κοινέ θέσεις που όπως είπα και στην αρχή θα ήθελα να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερη αυτή η συνένεση για να ενισχυθεί ακριβώς και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την τόσο κεφαλαιόδη φάση τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά ήθελα να πω και είμαι έτοιμη να απαντήσω στα ερωτήματα Σα Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φεραίρα. Εκ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, ο κύριο Γκοζές. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αναγκάστηκα να εγκαταλείψω την αίθουσα για λίγο, αλλά παρόλα αυτά διάβασα προσεκτικά την έκθεση και επομένως μπορώ να τη σχολιάσω. Μπορώ να πω ότι το κείμενο αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από το ΕΛΚΕ στην παρούσα του μορφή, διότι απομακρύνεται εντελώς από τις συμβαστικές λύσεις τις οποίες είχαμε βρει στο, για το προηγούμενο κείμενο όσον αφορά το εξάμεινο και επομένως δεν είναι δυνατόν, δεν μου φαίνεται καθόλου λογικό από τη μια χρονιά στην άλλη να αλλάξουμε ριζικά θέση. Έχουμε καταθέσει ε, σειρά τροπολογιών μέσω ε, και της κυρίας Βαρτμαντ Κόλ ε, και του συναδέλφου Λάγκερ και βεβαίως είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συζήτηση ε, αυτή είναι η θέση μου άλλωστε όσον αφορά όλα τα ζητήματα, δηλαδή προσπάθεια εξέβρεσης συμβιβαστικών λύσεων με την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν φάσκουμε και αντιφάσκουμε. Ε, και να μην αναιρούνται τα αποτελέσματα των συμβιβασμών ε, που βεβαίως ήταν συμβιβασμοί από κάθε πλευρά και υποχωρήσεις από κάθε πλευρά. Η έκθεση κατά την άποψή μας απομακρύνεται πολύ από το πνεύμα ε, των συμφωνιών που είχαμε κάνει και των συμβασμών που είχαμε βρει. Και επομένως, όπως είπα και εξ αρχής, δεν θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε ε, την ε, έννοια της έκθεσης, την κατεύθυνση της έκθεσης. Ε, εμείς θέλουμε να στηρίξουμε την ε, Κομισιόν στην προσπάθειά της ε, να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στην εξυγίανση των οικονομικών, να προχωρήσουν και να συνεχίσουν τις διαφορετικές αλλαγές και να προσθέσουν και μέτρα υπέρ της ανάπτυξης. Νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσει πλέον αυτή η χονδροειδής αντιμετώπιση η οποία λέει λέει ότι ε, μονάχα οι πολιτικές ανάπτυξης ε, θα δώσουν ε, καλά αποτελέσματα, ενώ από την άλλη πλευρά λιτότητα και σφίξιμο του ζωναριού και επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό που ισχύει είναι ότι για να υπάρξει μια, ένα γερό οικοδόμημα θα πρέπει τα θεμέλια του να είναι γερά. Επομένως θέση μας είναι αυτή της συμφιλίωσης μεταξύ αφενός της ανάγκης ε, σταθεροποίησης ε, και εξυγίανσης των οικονομικών ε, με από την άλλη πλευρά μέτρα τα οποία θα εντείνουν και θα βοηθούν την ανάπτυξη και με τον τρόπο αυτό θα επιτύχουμε τη μείωση του χρέους αλλά και την πρόληψη μελλοντικών οικονομικών κρίσεων που βεβαίως δεν θα αποφευθούν εάν δεν καταφέρουμε να έχουμε σαφείς οικονομικούς κανόνες. Κατά αυτή την έννοια θα είναι και πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον κύριο Γιούγκερ γιατί από τη μία πλευρά η κυρία Μέρκελ ε, στις ε, προβλέψεις του 2000 ε, και από την άλλη πλευρά ο κύριος Ολάντ μου δίνουν την αίσθηση ότι μιλάμε ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα αλλά με διαφορετικούς ε, τρόπους. Είναι σαν το κάθε μου αυτή να ακούει κάτι διαφορετικό. Ε, ε, και κατά αυτή την έννοια δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτούς τους οικονομικούς πολλαπλασιαστές που εισάγει η συγγήτρια και οι, οποία, και οι οποίοι αποσυντονίζουν την συζήτηση για τους σοσιαλιστές συναδέλφους ο πολλαπλασιαστής ε, έχει σαν ε, αποτέλεσμα ένα ευρώ στα δημόσια, στις δημόσιες δαπάνες μπορεί να γεννήσει παραπάνω από ένα ευρώ. Αυτό θα ήταν θαυμάσιο, θα ήταν τέλειο, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Ε, και ένα, εμείς φοβούμαστε ότι το ένα ευρώ των δημοσίων δαπανών μπορεί να μην είναι καν ισότιμο με ένα ευρώ. Από την άλλη πλευρά για να υπάρξουν δαπάνες πρέπει να υπάρξουν έσοδα, θα πρέπει να γεννηθούν, να δημιουργηθούν έσοδα ε, και ε, επομένως θα πρέπει αυτό να γίνει είτε ε, με την εισρωή νέων εσόδων είτε με το γνωστό, τη γνωστή επιστροφή των χρεών και επαναδανισμό που βεβαίως αυτό έχει και συγκεκριμένο κόστος. Απ' την άλλη πλευρά βεβαίως είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση και σε περαιτέρω συμβιβασμού, γιατί άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να βρεθούν ρεαλιστικές λύσεις και προτάσεις οι οποίες δεν θα μας δίνουν απλώς την αίσθηση αίσθηση ότι μπορούμε να φύγουμε από την ε, ε, κρίση, αλλά την βεβαιότητα ότι σιγά σιγά βγαίνουμε από αυτή την κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γκοζέσε εξ ονόματος των φιλελευθέρων, ο κύριος Δεμπακιά ε. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την εισηγήτρια βέβαια για την εισαγωγή της. Πρέπει να σας πω πως ευθυγραμμίζομαι με αυτά που είπε το ΕΛΚ. Γιατί Πιστεύω και το έχετε δει με τις τόσο πολλές τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, ότι τουλάχιστον ορισμένοι από εμά πιστεύουμε ότι πηγαίνει πολύ μακριά αυτή η έκθεση και όχι προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν οι διαφορές δηλαδή που ανέφερε και η συγκήτρια, είναι πραγματικές, βασίζονται σε γεγονότα, πολλές από αυτές και σε ιδεολογία βέβαια. Τώρα πολλοί από τους συναδέρφους ε, έχουν να κάνουν σχόλια, αλλά για τα δύο σημεία κυρίως που ανέφερε η συγγήτρια, δηλαδή πρώτα απ' όλα πώς θα ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος του Κοινοβουλίου μας. Εδώ νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ συμφωνούμε. Αν βέβαια μιλάμε και για το ίδιο πράγμα, γιατί είναι πολύ βασικό να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Αλλά το Κοινοβούλιο από την άλλη μεριά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί τότε θα κάνουμε το ίδιο λάθο που έκανε και το Συμβούλιο κατά το παρελθόν. Δηλαδή ότι θα καθόμαστε μεταξύ μα θα συζητάμε και θα διαπραγματευόμαστε χωρίς όμως να καταφέρουμε να πετύχουμε μεταρρυθμίσει γιατί θέλουμε τη δέσμη των 6, των 6 μέτρων και το ευρωπαϊκό εξάμενο ακριβώ για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις. Σίγουρα η κρίση είναι πολύ σοβαρή και προτείνει ε, μέτρα για να αντικατασταθεί, μάλλον για να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή, για παράδειγμα η ανεργία των νέων. Εντάξει, αλλά όπως είπε και ο κύριος Γκοζές, δεν μπορούμε να τα ε, πετύχουμε ε, όλα αυτά με τον τρόπο που προτείνει η συγγήτρια. Η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά πρέπει να υπάρξει κάποια αισιοδοξία γιατί βλέπουμε ότι είναι κάπως καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από την κρίση. Και αυτά που συζητάμε, για παράδειγμα το δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή που είπε και ο κύριος Γκοζές, πράγματι έγιναν κάποια λάθη κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά να δούμε και όλα όσα λέει το IMF, το, Ευρωπαϊκό, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Εγώ βέβαια είμαι πρόσφατα εδώ, αλλά καλά θα κάνουμε να κοιτάμε και μακροπρόθεσμα τι θα γίνεται. Αν ε, βραχυπρόθεσμα ε, αλλάξουμε, δεν σημαίνει ότι μακροπρόθεσμα θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Η κρίση έχει επίσης καταδείξει ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να συνεχίζουν να χρεώνονται όπως έκαναν κατά το παρελθόν. Χρειαζόμαστε διαρθρωτικές αλλαγές, ε, χρειαζόμαστε περιορισμούς στις δαπάνες, άρα χρειάζονται μεταρρυθμίσεις πολύ γρήγορα και άρα εδώ υπάρχει περιθώριο και για συζητήσεις σε τεχνολογικό επίπεδο αλλά και σε ιδεολογικό. Είμαστε έτοιμοι εμείς και ανοιχτοί να συζητήσουμε για να πετύχουμε συμβιβασμούς όπως έχουμε κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν με το πακέτο των έξι νομοθετικών μέτρων ή και με το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ελπίζω έτσι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Τεβάκερ. Εκ μέρους των ε, Βρετανών Συντηρητικών δεν βλέπω κανέναν. Η κυρία Τούλνεμεν τότε έχει το λόγο εκ μέρους των Πρασίνων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που καθυστέρησα, γιατί ήμουν στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω την παρουσίαση της κυρίας Φερέιρα. Αυτό είναι το κακό με όλες αυτές τις επιτροπές. Δεν προφταίνουμε. <clears throat> Χαιρετίζουμε την έκθεση, αλλά βλέπουμε και κάποια ανάγκη να υπάρξουν βελτιώσεις και περιθώριο βελτιώσεων και θα ήθελα να πω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε, όπως αναφέρθηκε και από, το προηγου... από τους προηγούμενους ομιλητές, ότι υπάρχουν και κάποιες διαφορές προσέγγισης και γι' αυτό υπάρχουν τροπολογίες που κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Εμείς ως πράσινοι βέβαια θέλουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. και ξέρουμε ότι υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές που πρέπει κάπως να τις ξεπεράσουμε. Και στο παρελθόν είχαμε τέτοια προβλήματα, αλλά νομίζω έχουμε καταφέρει να τα υπερπηδήσουμε. Το ίδιο πρέπει να γίνει και τώρα. Τώρα κάποιο είπε ότι έχει τελειώσει η κρίση, δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. <clears throat> αυτό μου φάνηκε υπερβολικά αισιόδοξο. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι υπήρξε και κάποια πρόοδος αλλά θα πρέπει να δούμε και τις ανησυχητικές εξελίξεις οι οποίες παρατηρούνται. Παραδείγματος χάρη η συνεχώς ανερχόμενη ανεργία, η αύξηση του κρατικού χρέους και το γεγονός ότι δεν υπάρχει πραγματική ανάπτυξη εφέτος τουλάχιστον και μέσα στα επόμενα χρόνια, κάτι που είναι απαραίτητο για την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Κάτι ακόμα το οποίο θέλω να <clears throat> διερευνήσω με τους άλλους συζητητές είναι ότι κάπως υπάρχει μια πιο ισορροπημένη αντιμετώπιση ανεξάρτητα από διάφορες πολιτικές παρατάξεις. Υπήρξε η πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που τόνισε τον ε, αρνητικό χαρακτήρα της μείωσης των δημοσίων δαπανών σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, ότι ήταν πιο μεγάλο το αποτέλεσμα από ό,τι προσδοκόταν προηγουμένως Όλα αυτά δείχνουν ότι η εμπειρία και η γνώση η οποία έχει αποκτηθεί σε εμπειρικό επίπεδο είναι κάτι το οποίο πρέπει και αυτό να αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση μεταξύ των σκιωδών συγητών. Και τρία σημεία για τα οποία μπορούμε να βρούμε ίσως κάποια συμφωνία. Καταρχήν για τα δημόσια οικονομικά. Και εγώ είμαι νεόφερτη σε αυτή την επιτροπή. Από ό,τι έχω παρακολουθήσει και από ό,τι ξέρω από του άλλου συναδέλφου, υπήρχε πάντα μια συμφωνία μεταξύ των συναδέλφων <clears throat> να έχουμε μια αντιμετώπιση η οποία να είναι μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Και πήγε πάντα μια η συμφωνία να είμαστε επιφυλακτικοί σε σχέση με την προσθήκη νέων χρεών μέσα στη χώρα, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης θέλαμε να εισαγάγουμε μια ευκαμψία σε όλα αυτά τα θέματα όπως κάναμε στο Six και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτή τη δυνατότητα ευκαμψία σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά και στην τρέχουσα έκθεση. Ένα δεύτερο τώρα θέμα είναι το θέμα της δημοκρατικής λογοδοσίας που τονίζει η Επιτροπή μας πάντα. Έχουμε το νέο βαθμολόγιο της Κομισιόν, το οποίο το σεβόμαστε, αλλά δεν ακολουθούσε αυτό το οποίο είχε συμφωνηθεί στο παρελθόν να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στην εκπόνηση του. Αυτό είναι κάτι λοιπόν που πρέπει να το τονίσουμε και πάλι με στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Πρέπει να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και να γίνεται σεβαστή και η γνώμη του. Τρίτο σημείο, ανταγωνιστικότητα. <clears throat> Θα πρέπει να γνωρίσουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση. Το γεγονός ότι μειώνεται η ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης ότι βρισκόμαστε σε πίεση ως ε, περιοχή του κόσμου. Επομένως και εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους κινδύνους προς την ανταγωνιστικότητα και επομένως και προς την ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επίσης μας ενδιαφέρει η αποδοτική χρήση των πόρων που θα οδηγήσει και σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Αυτά λοιπόν προς το παρόν θα ήθελα να πω και εμείς έχουμε καταθέσει πολλές τροπολογίες, ίσως πάρα πολλές, περισσότερο από ό,τι πρέπει. Αλλά προσβλέπουμε στην περαιτέρω συζήτηση με την εισηγήτρια. Ας προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ κυρία Τούρουνεν. <coughs> Πάμε τώρα στην συζήτηση. Υπάρχουν δύο οι οποίοι ζήτησαν το λόγο. Α, συγγνώμη. Ο κύριος Κλούτε, εξ ονόματος της ε, Γκουε, δεν είχαμε το όνομά σας. Καταρχήν εσείς λοιπόν, <coughs> συγγνώμη, συγγνώμη κύριε Κλούτε. Ναι, η Μαρίζα Ματίας είναι υπεύθυνη για το θέμα αυτό. Εγώ ε, την αντικαστώ απλώς, μου ζήτησε να μεταφέρω μερικά α, στοιχεία από τη δική της θέση. Εγώ πιστεύω ότι καταρχήν υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά τα θέματα του προϋπολογισμού των κρατών μελών. Η κάθε ομάδα βέβαια έχει ένα διαφορετικό τρόπο να το αντιμετωπίσει αυτό. Θέλουμε να το δούμε μονάχα σε ό,τι αφορά τα θέματα της ε, χρέωσης του κρατικού χρέους ή θα πρέπει να δούμε και τη δομή του προϋπολογισμού. Υπάρχει κατά τη διάρκεια <clears throat> να θυμηθούμε ότι μέσα στα πλαίσια της κρίσης υπήρξαν πολλές χώρες οι οποίες χρησιμοποίησαν φορολογικά μέτρα για να αποτρέψουν μια διεύρυνση των, μια περαιτέρω ε, διεύρυνση των ε, ελλημάτων τους. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Και επίσης αν δούμε και τις ανισομέρειες οι οποίες υπάρχουν, σας υπενθυμίζω την έκθεση του Άντορ η οποία θα δημοσιευτεί αυτή τη βδομάδα, που είναι ο αρμόδιος επίτροπος για τα κοινωνικά θέματα, όπου καθιστά απόλυτα σαφές ότι υπάρχει μια αύξηση της ανισότητας και της ένδειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό υποστηρίζει τα λόγια της εισηγήτριας. Επανέρχομαι λοιπόν στην έκθεση της Ελίζα. Εμείς στο παρελθόν <clears throat> είχαμε σταθεί κάπως επικριτικοί για την ε, οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Η έκθεση της κυρίας Φερέιρα όμως βρίσκει σε μεγάλο βαθμό την υποστήριξή μας. Θεωρώ ότι αυτά τα οποία έχει παρουσιάσει η συγγήτρια είναι γενικά θετικά και ιδίως το γεγονός ότι τονίζει τις αρνητικές ε, επιπτώσεις της κρίσης, ιδίως την μεγαλύτερη κοινωνικο-οικονομική ανισότητα η οποία δημιουργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά τα υποστηρίζουμε. Επίσης, είναι σημαντικό αυτό που λέω ότι πρέπει να μειωθούν και οι ανισομέρειες στο εμπορικό ισοζύγιο. Ξέρετε ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας έχει ακόμα τεράστια πλεονάσματα και εξακολουθεί αυτό να αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Η Κομισιόν στις ε, εκθέσεις της το 2011 και το 2012 έχει ήδη αναφερθεί στο θέμα αυτό. Επίσης, οι συνέπειες των μέτρων λιτότητος και η μείωση της ζήτησης είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναφερθεί και επίσης το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετά, αρκετές θετικές οθήσεις για την ε, ανάπτυξη. Υποστηρίζουμε λοιπόν την ανάγκη να τονίσουμε το στόχο της ανάπτυξης. Πέραν λοιπόν της γενικής υποστήριξης που έχω στην έκθεση Φερέρα, που έχει μάλλον η κυρία Ματίας, υπάρχουν και ορισμένα σημεία κριτικής τα οποία θα ήθελα να αναφέρω, τα οποία ίσως οδηγήσουν σε βελτίωση της έκθεσης. Για μας θα έπρεπε να αναφέρετε πιο σαφές ότι η διαδικασία φιλελευθερωποίησης και απορρίθμισης των χρηματαγορών και χρηματοπιστωτικών αγορών έχει συμβάλει τα μάλα στην κρίση, και αυτή η πολιτική πρέπει να τροποποιηθεί κατεπηγόντως, αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο είναι εν εξέλιξη αυτή τη στιγμή, η αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά κατά τη δική μου άποψη αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει με πιο στεναρό τρόπο. Επίσης, η εισαγωγή του ευρώ και επίσης η από πληθωριστικού χαρακτήρα μισθολογική πολιτική μια συγκεκριμένη χώρα τη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Γερμανία έπαιξε και αυτή ρόλο στην ανάπτυξη τη κρίση, όπω αναγνώρισε η Κομισιόν στι συστάσει του 2012. Και επίση θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν πρόκειται για μία ή δύο χώρε οι οποίε πλήττονται από την κρίση, αλλά για όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όλου του πολίτε. Είναι μια κρίση που αρχίζει να την νιώθει ακόμα και η Γερμανία γιατί η δυνατότητα να δίδονται διέξοδες στις εξαγωγέ της Γερμανίας στην Νότια Ευρώπη έχει μειωθεί σε σημαντικό χαρακτήρα. Επίσης, <clears throat> ε, χρειάζεται μια μεγαλύτερη συμμετρικότητα γιατί αντιμετωπίζονται διαφορετικά τα πλεονάσματα από ότι τα ελλείμματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Χωρίς μια τέτοια αντιμετώπιση δεν μπορεί να είναι εφικτή η επίλυση του πρόβληματος. Επίσης ξέρουμε ότι δεν έχουν επιτύχει τα μέτρα παροχής ρευστότητος προς τις τράπεζες. Τα χρήματα αυτά έχουν ουσιαστικά συσσωρευτεί και αποθυσαυριστεί από τα πιστοτικά ιδρύματα, αλλά δεν καταλήγουν στην πραγματική οικονομία. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξουν προγράμματα τα οποία θα έχουν χαρακτήρα μακροοικονομικής εξισορρόψης, να υπάρξουν επίσης διαδικασίες για την αναδιάθρωση των χρεών και η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών είναι θέματα τα οποία για μας είναι απαραίτητα. Φυσικά όμως αυτό δεν πρέπει να γίνει αυτόνομα, αλλά πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με παροχή κινήτρων για ανάπτυξη. Ακόμα μία παρατήρηση δική μου πέραν αυτό της κυρίας Ματίας θα ήθελα να αναφέρω τώρα. Η Κομισιόν εστιάζει και στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναρωτιέμαι αν αυτό είναι μια καλή ε, προσέγγιση, αν με τον τρόπο αυτό δεν κατακαιρματίζεται ιδιαίτερα η αντιμετώπιση του προβλήματος μήπως θα είχε πιο πολύ νόημα να εστιάσει την προσοχή της η Κομισιόν στα πιο κέρια κράτη, σε αυτά τα οποία ε, εμφανίζονται τα πιο μεγάλα προβλήματα. Αν αυτό θα ήταν πιο λυσιτελές θα μας έδινε περισσότερα στοιχεία. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι μια πρόταση την οποία θα μπορούσε να συζητήσει κανείς. Αυτά ήθελα να πω λοιπόν και η ελπίδα μου είναι ότι δεν θα αποδυναμωθεί τόσο πολύ η έκθεση της κυρίας Φερέιρα μετά από την διαδικασία ε, συμβιβασμών. Ελπίζω ότι κάποια από τα βασικά στοιχεία της έκθεσης αυτής θα μπορέσουν να παραμείνουν και να έχουν στεναρό χαρακτήρα. Ευχαριστώ κύριε Κλούτε. Δίνω το λόγο στον κύριο Κλίντς. <clears throat> Σας ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ δύο-τρεις σύντομες παρατηρήσεις μόνο θα να κάνω γιατί ο Φίλιπ Ντεμπάκερ εξ όνομα της ομάδας μας έχει ήδη παρουσιάσει τη θέση μας. Η Ελίζα Φερέιρα έχει αναφέρει σε ένα παράρτημα τρεις θεματολογίες. Καταρχήν το θέμα της ε, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Δεύτερον το θέμα του δημοκρατικού ελέγχου και της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Και επίσης εξέτασε τα θέματα εναλλακτικών κατευθύνσεων πέραν της πολιτικής λιτότητος. Εγώ συμμερίζομαι την άποψη ότι η φοροδιαφυγή είναι μια εγκληματική δραστηριότητα και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η φοροαποφυγή τώρα, εφόσον χρησιμοποιεί τα νομικά παραθυράκια, είναι κάτι το οποίο οποιοδήποτε επικεφαλής των των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μιας επιχείρησης θα το χρησιμοποιήσει. Είναι η δουλειά του ουσιαστικά ενός ε, επικεφαλής επιχείρησης να βελτιστοποιήσει τις ευκαιρίες που του δίδονται για να μειωθεί η φορολογία του. Αυτό δεν πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε σαν αδίκημα. Απλώς θα πρέπει να τροποποιήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο τις ε, δικές μας ρυθμίσεις ώστε να μην αφήνουμε να υπάρχουν τέτοιου είδους παραθυράκια και δυνατότητες αποφύγης φορολογίας. Και εδώ υπάρχουν διάφορα στοιχεία, διάφορα σημεία τα οποία αναφέρει η κυρία Φερέρα. Εγώ όμως είμαι 9 χρόνια σε αυτό το κοινοβούλιο και δεν έχω δει καμία σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτό. Εδώ δεν μπορούμε να κλείσουμε τα παραθυράκια τα οποία οδηγούν σε μαζικές απάτες για τον φόρο προστιθέμενης αξίας, πόσο μάλλον να αντιμετωπίσουμε γενικότερα το θέμα αυτό. Δεύτερον, το θέμα του δημοκρατικού ελέγχου και του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εγώ υποστηρίζω αυτήν τη θέση. Θα πρέπει να σταθούμε στεναροί και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έρχομαι τώρα στις προτάσεις της Ελίζα για το πώ ε, αντί για μια πολιτική λιτότητα ή αυστηρότητα μπορούμε να ακολουθήσουμε μια διαφορετική πολιτική. Εγώ συμφωνώ με τον Ζαν Πολ. Στη δεκαετία του 1970 ξεκίνησε αυτή η πολιτική των κυβερνήσεων να δίδουν περισσότερες παροχές από ό,τι είχαν φορολογικά έσοδα. Στη χώρα μου υπήρξε αυτή η χρήση κενσιανών πολιτικών που είχε τότε πληθωρισμό 5% και 5% ανεργία όταν ξεκίνησε και τώρα θα ήμασταν ευτυχεί να έχουμε μόνο 5%, αλλά αυτή η πολιτική οδήγησε τελικά σε 10% πληθωρισμό, 10% ανεργία. Επομένω, αυτή η πολιτική δεν έχει αποδώσει. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πραγματική κρίση αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Εάν δεν υπάρξει αυτή η επαναφορά της εμπιστοσύνη και της αξιοπιστίας δεν μπορούμε να ξανααποδηθούμε σε μια διαδικασία δημιουργίας περαιτέρω χρεών. Και οι αγορές παρατηρούν τη διαδικασία εδραίωσης των δημοσιονομικών και δεν θα δεχτούν να χρηματοδοτήσουν τους εθνικούς, τα εθνικά ελλείμματα με επιτόκια χαμηλά. Δεν μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά με θεωρητικολογίες. Μόνο με εδραίωση των δημοσίων οικονομικών θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πόρους και δυνατότητες ανάπτυξης. Όλα αυτά απαιτούν μεγαλύτερη ορθολογικοποίηση και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Τα έχει τονίσει αυτά ο κύριος Μόντι ότι δεν έχει ακόμα συμπληρωθεί η εσωτερική αγορά, ιδίως σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες για τις ανισομέρειες επίσης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο <clears throat> θα πρέπει να το βλέπουμε σε τακτά διαστήματα. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις. Το να θεωρήσουμε ότι μπορούμε με μια κεντρική σχεδίαση, με μια κεντρική διαδικασία φορολογίας να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες, αυτό είναι μια ουτοπία μπορούμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιοι είναι οι λόγοι για αυτές τις ανισότητες και πού βρίσκονται τα προβλήματα. Πολλές φορές υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγικότητα σε ορισμένες χώρες από ό,τι σε άλλες ή αλλού είναι ισχυρότερο το εργασιακό κόστος από ό,τι σε άλλες χώρες και μπορούμε επομένω να πάρουμε κάποια μέτρα για όλα αυτά. Αλλά το να θεωρούμε ότι μπορούμε από τις Βρυξέλλες με κεντρικό τρόπο να μπορέσουμε στον διηνικές να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά για μένα είναι μια λαθασμένη αντίποση. Αυτό οδηγεί σε μια κεντρική σχεδίαση της Οικονομία τη αγορά, το οποίο εγώ το απορρίπτω. Τρίτον, για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εγώ συμφωνώ με την Ελίζα ότι υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίηση των κονδυλίων τη Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά έχοντα μιλήσει με το νέο πρόβλημα, της με το νέο πρόεδρο τη Επιτροπή, της Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων, το θέμα δεν είναι χρηματοδότηση. Μπορούμε να διευρύνουμε το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής τραπεζα Επενδύσεων και οι, όλες οι χώρες και οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συμμετάσχει σε αυτό. Αλλά αυτό δεν οδηγεί σε κάποια λύση. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αρκετά ελκυστικά προγράμματα στα οποία να επενδυθούν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και γι' αυτό πρέπει να γίνει μια έκκληση προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρουσιάσουν προγράμματα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν ε, από την Τράπεζα Επενδύσεων και τα οποία όμως συμπεριλαμβάνουν και κάποιο δυναμικό ανάπτυξης. Και τέλος, το θέμα της κερδοσκοπίας. Όλοι μας εκφράζουμε την αποστροφή μας για τις κερδοσκοπικές επιθέσεις κατά του ευρώ. Αν θέλουμε όμως να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν έρχονται στα καλακαθούμενα είναι απλώς επιθέσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τις αδυναμίες, εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες ορισμένων κρατών και των δημοσίων οικονομικών τους και είναι και απάβγασμα του γεγονότος ότι δεν είναι βιώσιμη η κατεύθυνση ορισμένων χωρών στον οικονομικό πεδίο. Έχουμε καταθέσει και πολλές προτάσεις για τις ε, υπηρεσίες πιστοληπτικής αξιολόγησης και εκεί θα μπορούσαν να υπάρξουν βέβαια βελτιώσεις, αλλά αυτό δεν μπορεί να, να αποτρέψει τελείως τις επιθέσεις. Ούτε είναι ο σωστός δρόμος να πούμε ότι θα απαγορεύεται να υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση του κρατικού χρέους. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει τις κερδοσκοπικές επιθέσεις. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκίγκολ έχει τώρα το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, Αρχικά δεν σκόπευα να πάρω το λόγο στη συζήτηση αυτή. Αλλά πρέπει να σας πω ότι έχω την αίσθηση ότι ορισμένοι νομίζουν ότι έχει ήδη ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Αυτό είναι θλιβερό. Έχουμε προβλήματα, πραγματικά, ουσιαστικά προβλήματα. Και η συζήτηση για την έκθεση αυτή, έτσι όπως την ακούω, αλλά και η ίδια η έκθεση, με κάνει να σκέφτομαι σκέφτομαι ότι ιδεολογικοποιούμε το θέμα. Δεν πρέπει όμως. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να κοιτάξουμε τα διάφορα θέματα ξεχωριστά. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ποια είναι η πραγματικότητα στις χώρες αυτές πρώτα απ' όλα. Είναι θλιβερή η συζήτηση. Έχω την εντύπωση ότι γενικά όταν μιλάμε για την ε, κρίση της Ευρωζώνης, κοιτάμε πάρα πολύ λίγο το πόσο υποφέρουν οι άνεργοι στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Αν δείτε τη νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό το δείχνει ξεκάθαρα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε λοιπόν πώς υποφέρει ο κόσμος εκεί. Δεύτερον, για τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές. Είναι, λες, και πρόκειται για μια σοσιαλιστική συνωμοσία. Δεν είναι όμως. Δεν είναι τέτοια θεωρία. Αν να διαβάσετε την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, φαίνεται ξεκάθαρα εκεί. Ήταν πολύ σημαντική η έκθεση αυτή. Γιατί, γιατί παραδέχτηκαν ότι έκαναν ε, λάθη στην κρίση τους και τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 ακριβώς για τα ίδια οικονομικά στοιχεία. Ότι αν δηλαδή μειώσει σε μια κρίση τις δαπάνες, τότε κινδυνεύεις να μπει σε ένα φαύλο κύκλο που επιδεινώνει την κατάσταση. Και το κάνουν σε περίοδο κρίσης, λες και δεν είναι σε κρίση. Μα οποιοδήποτε θέλει να εξετάσει σοβαρά τις λύσεις σε μια οικονομική κρίση, πρέπει να δει την ισορροπία στον οικονομικό κύκλο. Οι πολιτικοί όμως έχουν αποτύχει, δεν έχουν εφαρμόσει αυτή την πολιτική. Και αυτό είναι σφάλμα. Και είναι σφάλμα να πούμε τώρα ότι υπάρχουν αυτοί οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές. Και Ζαν Πολ με κάθε φιλία που μας διακρίνει. Βέβαια, αν μια χώρα δαπανίσει ένα ευρώ, μπορεί να δημιουργήσει περισσότερη ζήτηση. Οπότε ο πολλαπλασιαστής είναι περισσότερο από το ένα. Αυτό είναι ένα γεγονός. Συνεπώς, το θέμα το καυτό είναι πού πάνε οι δημοσιονομικές δαπάνες και η ιδεολογική συζήτηση για το επίπεδο των δαπανών δεν είναι σωστό, γιατί υπάρχουν χώρες που έχουν ε, υψηλές δημοσιονομικές ε, δαπάνες, που πετυχαίνουν όμως με τους πολλαπλασιαστές και άλλες που πετυχαίνουν πολύ λιγότερα με τις ίδιες δαπάνες. Και έχουμε να μάθουμε πολλά από τις σκανδιναβικές χώρες. Άλλες πάνε πολύ άσχημα, όπως και η δικιά μου. Μπορείτε να το διαβάσετε και αυτό στις εκθέσεις που δίνουν τα στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ, ας είμαστε ισορροπημένοι και να βασιζόμαστε σε γεγονότα και όχι στην ιδεολογία μας. Το άλλο τώρα που θέλω να αναφέρω είναι το θέμα των κοινωνικών επιπτώσεων από την φόρα αποφυγή και την διαφυγή. Με αγαπητοί φίλοι, με κάθε πάλι φιλία που μας δεκρίνει. Ποια είναι η αρχή της ε, οικονομίας της κοινωνικής αγοράς είναι ξεκάθαρο και από τη σχολή του Φράιμπουργκ, που είναι η φιλοσοφική βάση του κόμματός μας. Δεν ζητάει από τους επιχειρηματίες ή από άλλους, ακόμα και από τους καταναλωτές, να μεγιστοποιήσουν το ωφέλη τους. Αλλά Τρόπιο, Σάντε, όλοι αυτοί πιστεύαν ότι η οικονομικη φορείς δεν θέλουν να μεγιστοποιήσουν μόνο τα δικά τους ωφέλη, αλλά θέλουν να λυθούν υπόψη και ηθικές αξίες. Ένας φιλελεύθερος ζητάει από το κράτος μόνο να είναι υπεύθυνο. Μα κοινωνική ευθύνη, οικολογική ευθύνη είναι κάτι που αποτελεί υποχρέωση για όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους καταναλωτές. Φυσικά και υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν μπορείς να ζητήσεις από οποιονδήποτε επιχειρηματία να σκοτώσει την επιχείρησή του χάρη του ανταγωνισμού. Όχι, αλλά τα φορολογικά ωφέλη είναι θέμα ευθύνη του καθενός. Εγώ πιστεύω ότι με τις παρατηρήσεις αυτές που κάνουν οι φιλελεύθεροι κάνουν λάθος γιατί δεν βασίζονται στις αρχές που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη και όπου υπάρχει συνένεση ουσιαστικά. Αυτά είχα να σας πω και για την κατάσταση στη Γερμανία. Έπειτα, όποιος ζητάει εξισορρόπηση για τον σχεδιασμό της οικονομίας, και αυτό είναι το λογικό. Τι ζητάει ο πάει με την έκθεσή του και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ε, έκθεση κοινωνικών στοιχείων που έχουμε από χτες ζητάει εξισορρόπηση όσον αφορά το κοινό νόμισμα δεν ζητάει κεντρική διάσταση. Δεν ζητάει απορρίθμιση να γίνει πιο φτωχή η Γερμανία και οι χώρες της Νότιας Ευρώπης να γίνουν πλούσιες. Όχι. Λέει ότι υπάρχει πάντα σε κάποια νομισματική ένωση. Το έχετε και στη Γερμανία και στην Ελβετία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένε Πολιτείε παντού. Δηλαδή, αν κάποιες περιοχές έχουν υψηλή ανάπτυξη και άλλες χαμηλή, τότε υπάρχουν αυτόματοι σταθεροποιητέ στο σύστημα για να εξορροπήσει την κατάσταση, ώστε να μην έχει 50% ανεργία των νέων σε μια περιοχή και 8% σε κάποια άλλη. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλα τα μέτρα τα οποία θέλουν να βάλουν τέτοιους αυτόματους σταθεροποιητές, λέτε ότι θυμίζουν σχεδιασμένη οικονομία. Ε, όχι, είναι τραγικό να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Ας επανέλθουμε καλύτερα στο πνεύμα συμβιβασμών και ας ξεχάσουμε την προεκλογική εκστρατεία και τις ιδεολογικές συζητήσεις. Πρέπει να σας πω ότι συνολικά είμαι αρκετά απογοητευμένος και συγγνώμη αν τα είπα σωμά. ομά. σε ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκίγκολτ. Αν δεν υπάρχουν άλλοι που ζητούν το λόγο, επιτρέψτε μου, και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, επιτρέψτε μου να πω να κάνω κι εγώ κάποια σχόλια. Συνήθως δεν μου αρέσει από τη θέση του Πρόεδρου να το κάνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι επικίνδυνο, πιστεύω, να συζητάμε εδώ την δυνατότητα διατήρησης των προγραμμάτων ε, οικονομικής εξυγένσης. Είναι λιγάκι όπως συμβαίνει με το λάδι και τη βενζίνη σε ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, χωρίς λάδι ε, οξυδώνεται και δεν ε, καταστρέφεται ο κινητήρας και χωρίς βενζίνη δεν μπορεί να προχωρήσει το αυτοκίνητο. Άρα χρειάζονται και τα δύο για να πετύχουμε το στόχο μας. Αυτό που έχει νόημα να συζητήσουμε εδώ είναι με ποιο ρυθμό θα εφαρμόσουμε τα προγράμματα οικονομικής εξυγίανσης. Αυτό είναι που πρέπει να έχουμε μπροστά μας πιστεύω. Από την άλλη, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και με το θέμα των ε, δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών. Δεν πρέπει να δημιουργούμε ε, ψευδείς ελπίδες. Δεν είναι το ίδιο το αποτέλεσμα ενός τέτοιου πολλαπλασιαστή όταν μια χώρα έχει ε, μεγάλο χρέος 40% με ένα άλλο κράτος που έχει δημόσιο χρέος ακόμα περισσότερο, 90% παραπάνω από 100% οι συνέπειες των δημοσιονομικών αυτών πολλαπλασιαστών στη δεύτερη περίπτωση είναι μηδενική. Ας είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί και να μην δημιουργούμε προσδοκίες που είναι ψευδοπροσδοκίες ουσιαστικά στον κόσμο. Αυτά είχα να πω εγώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια στην κυρία Φερέιρα. Παρακαλώ κύριε Φερέιρα. Μερσή λέει κυρία Φερέιρα. Θα μιλήσω αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για τα σχόλια και τις ε, τροπολογίες. Αναγνωρίζω ότι ο φίλος μου, ο κύριος ε, Γκοζές, ήρθε με μεγάλη ενέργεια έτσι, μετά τα Χριστούγεννα και καλωσορίζω έτσι, αυτό το δυναμισμό του. Αλλά βέβαια θα έπρεπε να είχε ακούσει προσεκτικότερα αυτά που είπα πριν μιλήσει και ο εκείνος, γιατί ε, προφανώς είχε προετοιμάσει τα όσα είπε ε, πέρα από αυτά που ε, είπα εγώ και πέρα από την ε, πρόθεση του, της εισηγητρίας. Προφανώς ήθελε να ακουστούν αυτά που ήθελε να πει. Εν πάση περιπτώσει δικαίωμά του. Ο καθένας μπορεί να έχει διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του θέματος. Πρέπει να πω ότι εγώ θα προσπαθήσω περαιτέρω να ε, ε, εξεύρω συμβιβαστικές λύσεις, όπως είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση. Πέραν τούτου, ενδεχομένως μπορεί να μην καταφέρουμε να βρούμε συνένεση. Δυστυχώς αυτά έχει η ζωή. Ε, θα ήταν βεβαίως πολύ κρίμα γιατί δεν θα περάσει ένα ισχυρό μήνυμα και ο στόχος που θέλουμε να επιτύχουμε δεν θα επιτευχθεί. Ε, πέραν τούτου δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτή είναι η ζωή όπως είπαμε. Έτσι είναι η ζωή. Τώρα, όσον αφορά τις διευκρινήσεις ε, και τις παρεμβάσεις του κυρίου Κλίνζε, που μπήκε σε πολλές λεπτομέρειες του θέματος, ε, και τις παρατηρήσεις του κύριου Γκίγκορτ και της κυρίας Έμιλι Τούμαν που μπήκαν σε πολλές λεπτομέρειες. Ε, τέλος ε, και ο Παύλος Άλβα ανέφερε την ουσία της συζήτησής μας. Γιατί σε τούτο το κείμενο δεν θέτουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό σχετικά με το αν χρειάζεται εξυγίανση των οικονομικών ή όχι ή σχετικά με το ε, ε, αν χρειάζεται ή όχι ο έλεγχος του χρέους. Δεν είναι εκεί το ερώτημα. Το ερώτημα είναι διαφορετικό. Πρέπει να προχωρήσουμε με το ρυθμό εξυγίανσης τον οποίο υλοποιούμε τώρα ή μήπως θα πρέπει να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα της μέχρι τούδε διαδικασίας και επομένως ενδεχομένως να επιβραδυνθεί ο ρυθμός της εξυγίανσης και να ξαναδούμε κάποια νέα μέτρα. Αυτό είναι το μόνο που ε, ε, συζητούμε. Βεβαίως δεν συζητούμε άλλα θέμα όπως ε, η καταπολέμηση της απάτης ή η λογοδοσία κτλ οι χώρες και οι οικονομίες ε, οι οποίες ε, έκαναν ό,τι τους ζητήθηκε πρότειναν μέτρα τα οποία δημιούργησαν ηφεσιακό ε, ε, περιβάλλον που ε, δημιούργησε μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που είχε εξ αρχής ειδωθεί και από αυτό το οποίο θα έπρεπε θεωρητικώς να αντιμετωπίσουν τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για δημοκρατικούς πολλαπλασιαστές τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν είχαν κάποια προεξοφλούμενα αποτελέσματα ε, ε, και βεβαίως ε, θα προχωρούσαν, θα, είχαν σαν αποτέλεσμα μια επιβράδυνση της οικονομίας. Αυτή η επιβράδυνση όμως σε, μερικός σε μερικές οικονομίες πολλαπλασιάστηκε επί τρία και επί τέσσερα και επομένως επιβράδυνε την οικονομική ανάπτυξη και τα μέτρα αυτά έχουν τέτοια αλληλοσύνδεση μεταξύ τους που μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο ύφεση από τον οποίο δεν μπορούμε πλέον να βγούμε. Άσχετα της πολιτικής ατζέντα, άσχετα από όλα τα άλλα ζητήματα που μπορεί να έχει κανείς στο, στο μυαλό του, παρακαλώ να δούμε την καθαρή πραγματικότητα ότι η Ευρωζώνη βρίσκεται σε ύφεση και έχει ένα ποσοστό ενεργείας που υπερβαίνει το 11%. Επομένως, με καθαρό μυαλό και αντικειμενικότητα να δούμε μήπως το παρακάναμε, μήπως τελικά πρέπει να σταματήσουμε λίγο με τα μέτρα που έχουμε πάρει μέχρι τώρα για να δούμε λίγο την κατάσταση και να, να την αντιμετωπίσουμε με πιο παραγωγικό τρόπο. Εδώ η αντίθεση δεν είναι ιδεολογική. Δεν πρέπει να είναι ιδεολογική. Πριν από τέσσερα χρόνια όταν είπαμε ότι η συνταγή δεν ήταν η σωστή, υποφέραμε και υπέφεραν πολλές χώρες, αλλά τώρα, τώρα ε, πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Μια και βλέπουμε ότι τελικά ε, καταστρέφεται, αποδυναμώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, χάνουμε τον έλεγχο. Παρόλα αυτά εξακολουθούμε να προχωράμε με τον ίδιο ρυθμό και με τον ίδιο τρόπο. Εγώ βεβαίω θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου έτσι ώστε να προτείνω λογικέ και αντικειμενικέ συμβιβαστικέ ε, λύσει. Όπω είπε και ο Στεν Γκίγκολτ, ε, θα πρέπει ε, να δούμε ποια είναι τα μέτρα, να τα μελετήσουμε. να δούμε αν στις χώρες οι οποίες έκαναν αυτό που τους ζητήθηκε το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο ή όχι. Θα προσπαθήσω λοιπόν να βρω συμβιβασμού. Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώρια συμβιβαστικών λύσεων, εάν συμφωνήσουμε όλοι βεβαίως ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί σχετικά με τη δουλειά που κάνουμε και θα κάνουμε, ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα ε, ποσά, σε συγκεκριμένα μέτρα, σε συγκεκριμένα αποτελέσματα ε, τα οποία έχουν ε, δώσει τα μέτρα αυτά, να μην μπούμε σε άλλες λογικές, να το ζήτημα δεν είναι αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτό που προτείνει η Κομισιόν. Οι πολίτε μα δεν μα εκλέγουν για να πούμε τι θαυμάσια δουλειά κάνει η Κομισιόν και πόσο τη λατρεύουμε και την αγαπάμε. Δεν είναι ούτε και ο στόχο μου. Στόχο μου είναι ε, Μάλλον όχι, δεν θέλω να έρθω εδώ και να πω εγώ κέρδισα την ε, μάχη ή ότι ε, ε, συμφώνησαν όλοι μαζί μου κτλ. Το ζήτημα είναι να είμαστε σαφείς εάν ε, τους στόχους που έχουμε θέσει, αν μπορούμε να τους επιτύχουμε καλύτερα με άλλα μέτρα. Αυτά. Αυτή είναι η πρόταση που κάνω ως εισηγήτρια. Βεβαίως θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, κάθε δυνατή προσπάθεια, με μεγάλη ειλικρίνεια και μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε ε, να προσπαθήσω να ε, συγκλίνω, ας πούμε, επί των διαφόρων στοιχείων ε, που έχουμε συμφωνήσει. Αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να πετσοκόψουμε αυτά που θέλουμε να πούμε έτσι ώστε στο τέλος ε, αυτά που θα πούμε εν τέλει να μην συμβάλλουν καθόλου στην επίλυση του προβλήματος της Ευρωζώνης και της Ευρώπης. Η πρόταση που γίνεται ε, με τα τρία βασικά ε, στοιχεία τα οποία σαφώς αναφέρθηκαν κυρίως από τον κύριο Κλίντς που αφορούν και σχετική προσαρμογή του, του επιλεγέντος ε, δρόμου και νομίζω ότι θα πρέπει να παραθέσουμε εδώ το Διεθνές Ταμείο που λέει ότι ή τα αποτελέσματα τα οποία έχουν ε, ε, ε, επιτευχθεί δεν είναι τέτοια και θα πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρηθούν. Και η δημοσιονομική πολιτική είναι ένας από τους πολλούς τομείς που θα πρέπει να επαναθεωρηθούν έτσι ώστε να καθοριστούν τα απαραίτητα βήματα τα οποία θα πρέπει να πάρει η κάθε μεμονωμένη χώρα όσον αφορά την εξυγίαση των οικονομικών της. Μιλάμε για εξυγίαση οικονομικών θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, να μην έχουμε καμία ιδεολογική ή ιδεολειπτική ε, προσέγγιση, να δούμε ποια είναι τα μέτρα τα οποία προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε και ποιος ήταν ο πραγματικός τους αντίκτυπος γιατί ε, είναι γεγονός ότι η Κομισιόν ε, αναγκάστηκε να επιβραδύνει την, το δρόμο της προσαρμογής ε, γιατί συμπέρανε ότι αυτά που συνέβησαν στην Πορτογαλία ή την Ισπανία δεν μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ότι αυτή η αναπροσαρμογή δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί τόσο γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα κάνω αυτά που πρέπει να κάνω, αυτά που οφείλω να κάνω σαν εισηγήτρια. Θα προσπαθήσω να ε, ε, επιτύχω κοινέ συμφωνίες όπου αυτό είναι δυνατόν και θα δούμε μαζί με τους συναδέλφους ε, που μπορούμε να καταλήξουμε. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα συνένεσης, λυπούμε ειλικρινά, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικά. Και σαν οικονομολόγος και σαν εκπρόσωπος εκλεγμένη των πολιτών της χώρας μου, δεν μπορώ να εθελοτυφλήσω σε αυτή την οικονομική κατάσταση την οποία διανύουμε. Είναι και δεοντολογικό το πρόβλημα, είναι, αφορά την προσωπική μου ηθική αντιμετώπιση αντιμετώπιση ε, του ζητήματος. Δεν μπορώ δηλαδή εγώ ε, να επιτύχω μια τεχνητή συνένεση αγνοώντας ε, την πραγματικότητα και δεν είναι δυνατόν με δειλία και μεγάλη πολιτική υποκρισία να αντιμετωπίσουμε τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φερέιρα. Εδώ κλείνει η συζήτηση κανονικά, αλλά μας μένουν άλλα 20 λεπτά μέχρι να μπούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι ο διάλογος που θα έχουμε με τον πρόεδρο τη Eurogroup, τον κύριο Γιούγκερ. Θα δώσω το λόγο στον σκιώδη συγητή των ε, συντηρητικών, τον κύριο Έπινγκ, και μετά, κύριε Φεραίρε, εφόσον επιθυμείτε, θα σας δώσω και πάλι το λόγο, εφόσον ε, επιθυμείτε να σχολιάσετε. Ο κύριος Έπινγκ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που δείτε το, το λόγο και συγγνώμη που έχασα τη χρονοθυρίδα μου γιατί ήμουν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για να θέσω ερωτήματα στην κυρία Άσταν για την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση Ευρωπαϊκής Ένωση. Είδατε πόσε τροπολογίε έχουν κατατεθεί, κύριε Πρόεδρε, για την έκθεση της κυρίας Φεραίρο. Όλα αυτά δείχνουν ότι πολλοί συνάδελφοι <clears throat> νιώθουν ανικανοποίηση με την έκθεση της ε, δεν έχουμε δει ακόμα βέβαια πρώτα συμβασμού, γι' αυτό στέκομαι μονάχα σε τρία σημεία, τα οποία είναι σημαντικά για τη δική μου ομάδα. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αντίθετα από την, εισαγωγή, από την εισηγήτρια, στο να θεωρήσουμε ότι η μελέτη του ε, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστέ, θα πρέπει να μα οδηγήσει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ο ο κ. συντάκτη αυτή της ε, έκθεσης είπε ότι τα συμπεράσματα εξαρτώνται και από τις υποθέσεις που θα ακολουθήσει κανείς. Υπάρχουν επίσης άλλες εκθέσεις που δείχνουν ότι η δημοσιονομική ενθάρρυνση, η εκπαικτατική πολιτική μπορεί να μην βοηθήσει σε χώρες οι οποίες είναι υπερχρεωμένες, έχουν πολλά προβλήματα. Επομένως, για τις χώρες αυτές δεν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω χρέωσης και δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Σε σχέση με τις τροπολογίες άλλων πολιτικών ομάδων, εγώ είμαι αισιόδοξο ότι μπορούμε να απαλύνουμε λιγάκι το ύφο αυτή τη έκθεση. Και επίση χαίρομαι για το γεγονό ότι πολλοί συνάδελφοι ε, διαφωνούν με την ιδέα της συζήτριας να απλωθεί η δημοσιονομική ε, αναπροσαρμογή σε περισσότερα χρόνια. Αυτή είναι η βασική συνταγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τόσο μεγάλη ανεργία χρειάζονται πραγματικά οι διαφορετικέ αλλαγέ για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα για να είναι πιο ευέλικτε οι αγορέ εργασία. Αυτό είναι η πρώτη μα προτεραιότητα. Τέλο, τελευταίο και τρίτο, θεωρώ ότι αυτή η έκθεση μα δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία να επιστήσουμε την προσοχή όλων στην ενιαία αγορά σαν πηγή ανάπτυξη και θέσεων εργασία. Στην τροπολογία 223, εγώ τονίζω τη σημασία να υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών που θέλουν να ακολουθήσουν την αρχή χώρα προέλευση για την ε, οδηγία σε σχέση με τι υπηρεσίε. Περιμένω λοιπόν τι συμβαστικέ σα τροπολογίε, κυρία Φερέρα, και ελπίζω ότι μπορούμε σε επικοδομητικό πνεύμα να συνεχίσουμε, αλλά ξέρω ότι στην Επιτροπή μα υπάρχει μια όκληση απόψεως σε σχέση με το αρχικό σας κείμενο. Ευχαριστώ. Κυρία Φερέρα, θέλετε να πείτε κάτι. Σας ευχαριστώ. Μπορεί να σας εντυπωσιάσει κύριε Έπινγκ, αλλά έχω δει κάποιες από τις τροπολογίες που καταθέσατε και συμφωνώ με πολλά από αυτά τα οποία λέτε. Και επίσης συμφωνώ και πολλές με τις τροπολογίες του κυρίου Γκοζές. Για αυτά που αναφέρατε τώρα, ναι, πιστεύω ότι η εσωτερική αγορά θα πρέπει να ενισχυθεί δεν την τροπολογία ίσως είναι υπερβολικά λεπτομεριακή, αλλά συμφωνώ γι' αυτό με την ενιαία αγορά και αυτό ίσω εκφεύγει κάπου του πεδίου εφαρμογή τη δική μα έκθεση. Συμφωνώ όμω για την ενιαία αγορά ότι είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη για την ε, δημοσιονομική παροχή ε, κινήτρων. Δεν είναι αυτό το οποίο μα απασχολεί αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για το θέμα του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή βλέπουμε ότι τα μέτρα τα οποία είχαν ε, προταθεί είχαν σαν στόχο να οδηγήσουν σε μια μικρή ε, μείωση της ταχύτητας της οικονομίας και οδήγησαν σε σχεδόν υφεσιακές καταστάσεις σε πάρα πολλές χώρες. Είναι σημαντικό λοιπόν να συγκρίνετε τα προβλεπόμενα αποτελέσματα των προγραμμάτων σταθεροποίησης σε πολλές χώρες όπου Βλέπετε σε πολλές χώρες ότι προβλεπόταν θα τελείωνε αυτή η μείωση, η μείωση της ανάπτυξης και θα είχαμε μια πρώτη απαρχή ανάπτυξης και αυτές οι χώρες τώρα έχουν μια ύφεση 3% ή οτιδήποτε ή παραπάνω. Όλες αυτές οι χώρες λοιπόν που θρησκευτικά ακολούθησαν αυτά τα μέτρα έχουν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση ύφεση. Αυτό συζητάμε σήμερα γιατί αν έχετε λανθασμένες εκτιμήσεις όταν εφαρμόζεται περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και αυτό μειώνει την εγχώρια ζήτηση, αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί αν έχουμε κάνει λάθος για την εκτίμηση του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή, καταρακώνουμε ουσιαστικά την οικονομία. Έχουμε μία μείωση ανάπτυξη τρει-τέσσερι φορέ μεγαλύτερη και έχουμε πρόβλημα να ξαναξεκινήσουμε και να αναθερμάνουμε και πάλι την οικονομία. Σε περιπτώσεις κρίσης υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι ο δημοσιονομικός ε, πολλαπλασιαστής μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τις φυσιολογικές εποχές και αυτό λέει και η έκθεση του Δουνουτού. Τέτοια πράγματα λοιπόν πρέπει να τα συζητήσουμε. <clears throat> Συμφωνώ με κάποιες από τις τροπολογίες σας και καταγράφω τις προτάσεις σας για συμβαστικές τροπολογίες. Και εγώ θέλω να δεχθώ να ακούσω τις παρατηρήσεις σας Απλώς, όπως είπα προηγουμένως, υπάρχει η ανάγκη ως Κοινοβούλιο και ως Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή να αποδηθούμε σε μια σοβαρή ανάλυση της κατάστασης και αυτό είναι κέριο στην τωρινή συγκυρία στην Ευρωζώνη και πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα με πολύ σοβαρό τρόπο και να προσπαθήσουμε επομένω και εγώ θα προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ τα μάλα τη συνεισφορέ όλων των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φερέρα. Σα πεθυμίζω ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα είναι στην επόμενη συνεδρίασή μας του Ιανουαρίου και θα γίνει η συζήτηση και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια το Φεβρουάριο για να είμαστε έτοιμοι ενώπιον του Εαρινού Συμβουλίου Κορυφής. Κάνουμε λοιπόν ένα μικρό διάλειμμα μέχρι μια στιγμή ο κ. Κοζές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, όταν δεν λέμε τα ίδια που λένε και άλλοι, μα περνάνε για καθυστερημένου. Κοιτάξτε όμω, μετά τη σημερινή συζήτηση, εγώ δεν βλέπω πώ είναι δυνατόν στι 21 Ιανουαρίου μπορούμε να έχουμε συμβαστικέ τροπολογίε. Είμαστε ήδη 10 του μηνό. Έχουμε 11 μέρε στη διάθεσή μα για τι συμβαστικέ πρωτοβουλίε δεν έχουμε δει καμία μέχρι τώρα. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι λογικό γιατί είχαμε τι χριστουγεννιάτικε διακοπέ, αλλά πώ θα τα καταφέρουμε μέχρι τι 21. Εκ των προτέρων μπορούμε να ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πρόεδρο. Κύριε Κοζέ, η επόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα που θα μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε, γιατί η μόνη δυνατότητα που έχουμε είναι να ψηφίσουμε το Φεβρουάριο. Δεν είναι δυνατόν ε, να έχουμε στις Βρυξέλλες ολομέλειες, ε, όπως γνωρίζετε, λόγω της κατάστασης του κτηρίου, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε τόσο ελαστικοί στις ημερομηνίε. Ο μόνος τρόπος είναι πώς που έχουμε προκειμένου να είναι έτοιμη έκθεση πριν από το Συμβούλιο το ΕΑΡΙΝΟ, είναι στις 21 Ιανουαρίου να ψηφίσουμε εδώ και το Φεβρουάριο να πάει η έκθεση στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Η κυρία Τούριναν έχει ζητήσει το λόγο γι' αυτό. Ναι. Μια πρόταση έχω να κάνω, να τη σκεφτεί η συγκήτρια. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε μία ώρα. Μήπως να βρούμε δύο ώρες. Γιατί καταλαβαίνω αυτό που λέτε ότι πρέπει να προλάβουμε τις προθεσμίες. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει πράγματι να ψηφίσουμε, αλλά μήπως να προβλέψουμε την επόμενη εβδομάδα μια ώρα παραπάνω. Πρόεδρος, ναι, ευχαριστώ κυρία Τουρινέν. Μου λέει η γραμματεία ότι θα μπορέσουμε όντως να έχουμε δύο ώρες στη διάθεσή μας την επόμενη εβδομάδα για να δουλέψουμε παραπάνω και να προλάβουμε έτσι. Ωραία, αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, τότε διακόπτουμε για λίγα λεπτά. Πρόεδρε, διακόπτω κύριος Γκοζές, για την δέσμη των δύο μέτρων που ακόμα δεν έχει ξεμπλοκαριστεί, δώσαμε πολύ περισσότερο χρόνο. Είναι γελίο. Πρόεδρος. Κύριε Κοζές, κύριε αυτή είναι άλλη συζήτηση. Αν θέλετε, έχουμε λίγα λεπτά, μπορούμε να το συζητήσουμε. Αν κάποιος θέλει να απαντήσει σε αυτό, ευχαριστώ, να το συζητήσουμε. Κύριε Κοζές, η κυρία Μπέρες. Παρακαλώ κυρία Μπέρες. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να μπερδευτώ τώρα στη συζήτηση, αλλά κοιτάξτε, εδώ δεν είμαστε τόσο στο νομοθετικό. Ο Ζαν Κοζές το γνωρίζει, όπως και άλλα μέλη εδώ στην Επιτροπή μας, ότι περιοριζόμαστε από τις ημερομηνίε. Προσπαθούμε δηλαδή να μην είμαστε εκτός προθεσμιών, σε σχέση με τη συζήτηση στο Συμβούλιο. Και στο Συμβούλιο, αναμφίβολα, οι συζητήσεις είναι εξίσου έντονες για την ανταγωνιστικότητα και τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές. Η συζήτηση για την ε, ανάπτυξη στο Ερεινό Συμβούλιο θα καταλήξει σε συστάσεις αναχώρα. Και όλα αυτά μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα που γνωρίζουμε ότι περιορίζει πολύ το κοινοβούλιο μας. Αλλά εμείς έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να παρέμβουμε και άρα πρέπει να τηρήσουμε τις προθεσμίες. Η μόνη δυνατότητα που έχουμε είναι το Φεβρουάριο να αποφασίσουμε στην Ολομέλεια. Γιατί αυτό έχει να κάνει και με τις συνεδριάσεις που οργανώνουμε με τα εθνικά κοινοβούλια. Οπότε με εκπλήσει λιγάκι η αντίδραση. Η δυσκολία δηλαδή αυτή που βρίσκουμε με το χρονοδιάγραμμα. Δεν είναι νομοθετικό το κείμενο, επαναλαμβάνω. Κύριε Γκοζές, ναι, πρόεδρε, κοιτάξτε. Με εκπλήσει η έκπληξη της εκπεπληγμένης κυρίας ε, Μπερές. Να δούμε ποιο ήταν το χρονοδιάγραμμα για τις συμβαστικές τροπολογίες στο προηγούμενο εξάμεινο. Ήμουνα εισηγητής. Πόσες συνεδριάσεις κάναμε. Πόσες συνεδριάσεις εργασίε για να καταλήξουμε στις συμβαστικές λύσεις. Πάνω από δέκα μέρες σίγουρα. Δεν τα έχω καταγράψει όλα αυτά γιατί δεν θεωρούσα ότι αυτό ήταν θεμελιώδους χαρακτήρα, αλλά μπορώ να ελέγξω Έκανα μια πρώτη συνάντηση με τους σκιώδεις, μετά ζήτησα από τους σκιώδεις ηγητές αν μπορούσα να συμπεριλάβω τις ιδέες τους για να καταλήξω στην τελική έκθεση. Έκανα μια προέκθεση, έβαλα τις ιδέες τους, είχα τροπολογίες πάνω σε αυτό το πρώτο σχέδιο, μετά συζητήσαμε τις τροπολογίες συμβασμού, δεν θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω αν οι συνεργάτες μου μπορούν να μου πούν πόσο κράτησαν αυτές οι διαπραγματεύσεις, αλλά χρειαστήκαμε πάνω από 10 μέρες για να βρούμε μια συμβαστική θέση. Αν ο στόχος είναι να δείξουμε ενώπιον των εκλογών ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διχασμένο, ας το κάνουμε έτσι. Αλλά αυτό θα αποδυναμώσει και τη θέση του Κοινοβουλίου και τη θέση μας για άλλα θέματα επίσης. Εγώ θα δώσω λοιπόν <clears throat> στη γραμματεία τα στοιχεία του χρονοδιαγράμματος το προηγούμενο εξάμεινο που οδήγησαν σε καλέ συμβαστικέ λύσει. Για μια καλή συμβαστική λύση χρειαζόμαστε χρόνο. Αν μας λένε τώρα δεχτείτε το ή απορρίψτε το, ξέρετε ποια θα είναι η θέση μα. Ε, ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρο. Κατανοώ ότι για το Τούπακ έχουν τελειώσει διαπραγματεύσεις και περιμένουμε μονάχα από ορισμένες πολιτικές ομάδες να έχουμε την απάντησή τους. Λοιπόν, η γραμματεία θα καταγράψει αυτά τα στοιχεία που θα τις δώσει ο κύριος Κώστα σχετικά. Ας κλείσουμε εδώ τη συζήτηση και περιμένουμε λίγα λεπτά μέχρι τις 11 ώστε να γίνει η συζήτηση με τον πρόεδρο της Ευρωομάδας, τον κύριο Γιούγκερ που όπως ξέρετε αυτή θα είναι η τελευταία συνάντηση που θα έχουμε με τον κύριο Γιούγκερ υπό την ιδιότητα αυτή του Πρόεδρου της Ευρωομάδας, του Γκρουπ. Ευχαριστώ όλους. Non, mais je suppose que c'était... Buon anno. Buon Ok. Obrigado. Okay, anybody else coming to shake hands? Just, just, just let's finish. Θέλετε να κάνετε και άλλες χειραψίες, σας τελειώνουμε αν μπορούμε, λέει η Πρόεδρος. me, um, ε, Πολύ μεγάλη χαρά για μένα να περάσουμε στο σημείο 6 της τη διάταξη, στον οικονομικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων με τον Jean-Claude Juncker, τον πρόεδρο της Ευρωομάδας. Είναι τμήμα των τακτικών ανταλλαγών απόψεων που έχουν θεσπιστεί μαζί με τον ε, Jean-Claude. Βέβαια όλα αυτά γίνονται σε πιο επίσημο επίπεδο μέσα στα πλαίσια του οικονομικού διαλόγου που προβλέπεται από το ΣΥΚΣΠΑΚ για τον ε, διάλογο με τον πρόεδρο της Ευρωομάδες. Όλα αυτά λοιπόν έχουν καθιερωθεί πια και σε επίσημο ε, επίπεδο. Η επιστολή μου <clears throat> της 26ης Ιουλίου πρότεινε μία επίσημη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωομάδος δύο φορέ το χρόνο, τον Ιανουάριο καταρχήν για να παρουσιαστεί το ετήσιο πρόγραμμα εργασία τη Ευρωομάδος και δεύτερον τον ε, Σεπτέμβριο για μια ενδιάμεση ε, εξέταση του ετήσιου προγράμματος και για την αντιμετώπιση των συστάσεων αναχώρα που θα είχε εγκρίνει το Συμβούλιο τον Ιούλιο. Και στην απάντησή σας εκφράσατε την θέλησή σας να έρχεστε ενώπιον της Επιτροπής μας δύο φορές το χρόνο μια φορά το, στην αρχή του χρόνου και μια φορά το φθινόπωρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Έχω επίγνωση του γεγονότος ότι έχετε σταθεί πρόεδρος της Ευρωομάδας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, 7 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για το έργο που έχετε φέρει σε πέρας και για την διαθεσιμότητά σας πάντα να έρχεστε ενώπιον της Επιτροπής σας, Επιτροπής μας, και ελπίζω και ο διάδοχός σας θα τηρήσει όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει έναντι της Επιτροπής μας και εξ ονοματός του πια. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ και προσβλέπουμε στην παρουσίασή σας. Περιμένουμε μια παρουσίαση 10-15 λεπτών <clears throat> σε σχέση με το έργο της Ευρωομάδας και τις ε, τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στις χώρες που βρίσκονται σε προγράμματα σταθεροποίησης και να περάσουμε μετά σε ομαδοποίησεις ομάδων ερωτήσεων και απαντήσεων μέσα σε πέντε λεπτά. Το σύστημα λοιπόν θα είναι <clears throat> ότι η ερώτηση και οι απάντηση θα πρέπει να καλύπτουν πέντε λεπτά το maximum. Εάν μιλήσει για πέντε λεπτά ο βουλευτής, εσείς δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Και με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε μια δυναμική ανταλλαγή απόψεων και ο στόχος είναι όλοι να μπορέσουν να περιοριστούν και να αποδεχθούν αυτό το πλαίσιο. <clears throat> Σας δίνω λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι λεπτομέρειες. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί φίλοι, γιατί έτσι πρέπει να απευθυνθώ σε πολλούς από εσά. Είμαι ενώπιον σας για τελευταία φορά ως πρόεδρος της Ευρωομάδος. Αλλά δεν πρόκειται τώρα να περάσουμε σε νοσταλγικές ε, ενθυμίσεις. Είναι χρόνος περισσότερο δράσης νοσταλγίας. το 2012 σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα για τη ζώνη του ευρώ. Ήταν σχετικά καλή χρονιά. και φυσικά εύχομαι καλή χρονιά για το 2013 σε όλους σας. Το 2012 πήραμε αποφάσεις οι οποίες είχαν σημαντικό και μακρόπνο χαρακτήρα. Έχουμε σταθεροποιήσει τη ζώνη του ευρώ. Και αν θυμηθείτε ότι το 2012, τον Ιανουάριο του 2012, πριν από ένα χρόνο, πολλοί από αυτούς που μας παρατηρούσαν και ακόμα και μερικοί από εμά τους ίδιους θεωρούσαν ότι η ζώνη του ευρώ πήγαινε κατευθείαν προς την καταστροφή, προς τη χρεοκοπία. Ιδίω στον αγγλοσαξονικό κόσμο υπήρξαν πολλοί εκτιμητές και αναλυτές που θεωρούσαν ότι κινδυνεύει να χαθεί, να καταστραφεί η ζώνη του ευρώ μέσα στο 2012, διαπίστωσαν ότι είναι ακόμα <clears throat> ζωντανή η ζώνη του ευρώ ότι η Ελλάδα την οποία προβλέπανε ότι θα αποχωρήσει από τη ζώνη του ευρώ βρίσκεται μέσα στη ζώνη του ευρώ ακόμα και βρίσκεται σε μια πορεία μεταρρυθμίσεων και αναπροσαρμογής από λοιπόν τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίησης <clears throat> με τα σχέδια σταθερότητας μια έκφραση που δεν μου αρέσει ιδιαίτερα για την Ελλάδα μετά από την ε, από το Δημοσιονομικό Σύμφωνο αφού καταφέραμε να βρούμε κάποιες λύσεις για τον Ισπανικό τραπεζικό τομέα. Μπορούμε να πούμε ότι σήμερα, τον Ιανουάριο του 2013, βρισκόμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που είχαμε να αντιμετωπίσουμε στην αρχή του 2012. η μέθοδος την οποία ακολούθησα ως επικεφαλής του, της Ευρωομάδος, του Eurogroup, ήταν και τώρα βέβαια κάνω ένα είδος απολογισμού. Ήταν μια ανάμιξη μιας ε, περιεκτικής μεθόδου, που είναι αυτή την οποία εγώ υποστηρίζω πάλι και η οποία βέβαια δεν μπορεί να περιλάβει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ο στόχος είναι να έχουμε μια περιεκτική αντιμετώπιση. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται να μπορούμε να παρακολουθούμε τις ε, επιδιώξεις και τις προσδοκίες των μεν και των δε. <clears throat> Και επίσης οι χώρες οι οποίες δεν είναι μέσα στη ζώνη του ευρώ, δεν θα πρέπει να αισθάνονται ότι είναι τα χαμένα παιδιά, τα αποπέδια του ευρώ κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό θέλησα πάντα να έχω μια περιεκτική προσέγγιση. Και αυτή η περιεκτική προσέγγιση φυσικά έχει και τα μειονεκτήματά της, έχει την απώλεια χρόνου που προκύπτει. Όταν πρέπει κανείς να απαντάει σε όλα τα τηλεφωνήματα, σε όλες τις αιτήσει που γίνονται προς την κατεύθυνσή του, Και αυτό ενώ οι συνεδριάσεις της Ευρωομάδος <clears throat> είναι μακροσκελής, πολλές φορές φτάνουν μέχρι τις πρωινές ώρες. Εγώ θέλω το ευρώ επειδή είναι το κοινό μας νόμισμα και επειδή είναι το νόμισμα όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνητικά, θέλω να εξασφαλίσω ότι όλοι θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν το λόγο αν δούμε το πόσο μέτρια ήταν τα αποτελέσματα που βγήκαν από πολλές συνεδριάσεις μας, θα μπορούσαμε να είχαμε ξεπερδέψει σε δυο 3 ώρες, αν δεν δίναμε το λόγο σε όλους. Και λέω ότι ίσως ο διάδοχός μου θα πρέπει να σκεφτεί περισσότερο για τα θέματα αυτά και ίσως να σκεφτεί ότι ναι, αυτά μπορούν να γίνονται πολύ πιο σύντομα. Πράγματι μπορούν να γίνουν όλα αυτά πολύ πιο σύντομα, αλλά θα δείτε μέσα σε έξι μήνες τι θα προκύψει εάν δεν δώσετε το χρόνο να ακούσετε όλες τις απόψεις σε επίπεδο ισότητας. Και τις χώρες που είναι στη ζώνη του ευρώ και τις χώρες που δεν είναι στη ζώνη του ευρώ. Νομίζω ότι μπορέσαμε το 2012 να εγκρίνουμε την Ευρωπαϊκή <clears throat> Δημοσιονομική Συνθήκη, η οποία ετέθη σε εφαρμογή μετά από την υπογραφή της από 12, από τουλάχιστον 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραμένουν κάποιες χώρες οι οποίες δεν έχουν ακόμα υπογράψει, δεν έχουν μάλλον κυρώσει αυτή την συμφωνία, όπως είναι το Βέλιο, όπως είναι οι κάτω χώρες και το Λουξεμβούργο, πρέπει να υπενθυμίσω. Η κύρωση αυτής της συνθήκης δεν είναι απόλυτα εξασφαλισμένη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, δεν έχει καμία επίπτωση, διότι, όπως σας είπα, έχει τεθεί σε εφαρμογή αυτή η συνθήκη. Και για το Λουξεμβούργο και μπορώ να μιλήσω και με το, σε εθνικό επίπεδο. Ξέρουμε ότι οι πράσινοι δεν θα υποστηρίξουν αυτή την ε, συνθήκη, γιατί θεωρούν μια συνθήκη γερμανικής έμπνευσης. Ότι είναι μια, κατά κάποιο τρόπο, ένα γερμανικό δικτάτ, μια γερμανική επιβολή. Είναι μια άποψη την οποία έχουν ορισμένοι ε, συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου. Εμείς χρειαζόμαστε να επιτύχουμε μια συνταγματικού χαρακτήρα πλειοψηφία δύο τρίτων για να γίνει η κύρωση αυτής της συμφωνίας. Επομένως και ευρύτερη συνένεση από αυτή του κυβερνητικού συνασπισμού και ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν σε άλλες χώρες. Ένα από τα βασικά προβλήματα επίσης είναι να βρούμε την απαραίτητη αρχή που απαιτεί αυτή η δημοσιονομική συνθήκη για την εποπτεία και την ε, <clears throat> εκτίμηση και τη σωστή διαχείριση των θεμάτων προϋπολογισμού στις μικρές χώρες. Γιατί για το Λουξεμβούργο να μπορέσει κανείς να φτιάξει μια νέα ανεξάρτητη αρχή δεν είναι απόλυτα αδύνατο, αλλά δεν είναι και εύκολο στα μεγάλα κράτη-μέλη, έχετε παντού εμπειρογνώμονες, έχετε άτομα τα οποία έχουν δείξει την αξία τους στις αναλύσεις τις οικονομικές που έχουν κάνει. Για ένα μικρό κράτος βέβαια αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο πολύπλοκο. Πίστευω θα τα καταφέρουμε παρόλα αυτά για τον Ευρωπαϊκό τώρα Μηχανισμό σταθερό... Σταθερότητος και είμαι ακόμα για τέσσερις μέρες ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμφώνου του Συστήματος Σταθερότητος έχουν δημιουργηθεί μηχανισμοί εδώ και 14 μήνες. Καταφέραμε λοιπόν να δημιουργήσουμε όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς, τώρα θα πρέπει να φροντίσουμε αυτοί οι μηχανισμοί να μπορέσουν να εκπληρώσουν όλες τις λειτουργίες οι οποίες τους έχουν αποδοθεί και αυτό περιλαμβάνει φυσικά και την άμεση ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Όταν λοιπόν έχει δημιουργηθεί η ενιαία εποπτική αρχή, θα χρειαστεί και μια συμφωνία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου προς τούτο. Είχαμε πει ότι θα δεχτούμε την ιδέα ότι η επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μπορεί να γίνεται από το ESM, από τον μηχανισμό σταθερότητος, τον οποίο έχουμε ήδη δημιουργήσει. Για το θέμα αυτό παραμένει βέβαια ένα μεγάλο ερωτηματικό σε σχέση με το κληροδότημα ή πιν του παρελθόντος. Μπορεί το, ο μηχανισμός σταθερότητος να δράσει και αναδρομικά να αντιμετωπίσει καταστάσεις που προϋπάρχουν του συστήματος σταθερότητας ή θα πρέπει να περιοριστεί η λειτουργία του στα νέα προβλήματα τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν στο μέλλον. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι χρειάζεται και κάποια αναδρομικότητα στη λειτουργία του μηχανισμού σταθερότητας, γιατί αλλιώς θα χάσει ένα μεγάλο μέρος από το νόημά του. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αναζητήσουμε κατά ανάγκη αιτίες και υπετίους για την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί. Για μένα όμως προέχει να χρησιμοποιηθεί και να είναι λειτουργικό αυτό το σύστημα σαν ε, θήκη εργαλείων κατά κάποιο τρόπο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Φυσικά όλα αυτά πρέπει να αποφασιστούν με ομοφωνία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου του Συστήματος Σταθερότητος και νομίζω ότι θα μπορέσουμε μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2013 να ακούσουμε όλες τις απόψεις και να καταλήξουμε σε κάποια θέση για τα θέματα αυτά. Έχουμε επίσης την έκθεση Φαν στην οποία έχω συμβάλει και εγώ, προσεκλήθη και εγώ να συμβάλλω. Όπως θυμάστε, σας το ξαναλέω για να έχει καταγραφεί ότι στην αρχή ήταν μια κοινή έκθεση των τεσσάρων προέδρων και κάποιοι από εσά την χαρακτήρισαν ως έκθεση σοφών. Εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες για τον επιστημονικό χαρακτήρα αυτής της ε, ονομασία σοφών και η για το επιστημονικό χαρακτήρα της έκθεσης και ιδίως για τον χαρακτηρισμό ορισμένων από εμά ως σοφών. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτή η έκθεση, η οποία έχει γίνει δεκτή, όχι απόλυτα στο σύνολό της από τον πρόεδρο Φαν Ρομπάι και τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν μετά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν και το είπα ανοιχτά, ήταν απογοητευτικά. Πολλές φορές ξεχνάμε ότι θα πρέπει όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά να έχουμε και κάποιο οδικό, οδικό χάρτη. Προς τα πού θέλουμε να πάει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Τι είναι η αλληλεγγύη μέσα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Πώς θα συνεργαστούμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε τους εταίρους μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Πώς θα χαράξουμε το μέλλον στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αντιμετωπίσαμε θέματα που είναι τελείως βραχυπρόθεσμα. Υπήρξε <clears throat> ακόμα μια ασάφεια για το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε την επόμενη δεκαετία για τα θέματα αυτά. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, ο κύριος Φαν Ρομπέι, έχει επιφορτιστεί μέχρι τις 6 Ιουνίου να παρουσιάσει ένα σύνολο ιδεών που θα ήθελα και εγώ να είναι καινοτόμε ιδέες σε σχέση με την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Οι ιδέες αυτές θα πρέπει να εκπονηθούν από τον κύριο Φανρομπάη μαζί με τον πρόεδρο της Κομισιόν. Βλέπετε ότι και το, η Ευρωομάδα δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον σε αυτή την ομάδα προβληματισμού για κάποιους λόγους. όλα αυτά θα πρέπει να οδηγήσουν σε κάποια διαβούλευση εξάντε για τα ζητήματα οικονομικής πολιτικής. Είναι χρήσιμο να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια για τα θέματα αυτά. Από το 1997 μιλάμε για την ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Μαζί με τον Ρομπέρ είχαμε προοδρεύσει σε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είχαμε καταφέρει να υπάρξει μια απόφαση των Υπουργών Οικονομικών εκείνη τη εποχή, όπου είπαμε να ενισχυθεί ο συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε σε ένα σύστημα όπου έχουμε μια όλο και πιο ισχυρή νομισματική ένωση, ενώ υστερεί και μένει πίσω η οικονομική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και 15 χρόνια, από το 1997, συζητάμε για το θέμα αυτό αυτοί οι οποίοι είχαν δισταγμούς και δεν θέλαν τότε να προχωρήσουν σε συντονισμό, είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα ζητούν επίμονα να γίνει αυτός ο συντονισμός. Δεν θέλω να μιλήσω για μια χώρα η οποία είναι ε, κοντά στο Λουξεμβούργο, ούτε για ένα βασίλειο το οποίο δεν απέχει μακριά από το Λουξεμβούργο. Καλώς ήλθατε λοιπόν στη λέση μας, αλλά τώρα θα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν μια κυβέρνηση θέλει να κάνει κάποια μεταρρύθμιση, κάποια διαρθρωτικού χαρακτήρα, θα πρέπει να παρουσιάζεται αυτή στην Ευρωομάδα. Και να μας εξηγήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί περί τίνος πρόκειται. Και να μπορούν και οι ομόλογοι του υπουργού, Υπουργοί να πούν πώς αυτό θα επηρεάσει τις δικές τους εθνικές πολιτικές για τα οικονομικά θέματα. Όλα αυτά θα είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση πιστεύω. Θα υπάρχουν ίσως πολλές επίσημες δηλώσεις. Αλλά η πραγματική υλοποίηση θα είναι ίσως πιο ισχνή. Τουλάχιστον όμως θα έχουμε κάποια κείμενα τα οποία θα μας επιτρέπουν να θέτουμε ερωτήματα μεταξύ μας μέσα στο, στην Ευρωομάδα. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. δεν θα ήθελα να εξαφανιστεί η κοινωνική μνήα και από την εκθέση του κυρίου Φαν Ρομπάη για το θέμα της κοινωνικής διάστασης Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Είναι πεποίθησή μου ότι είναι μια αναγκαιότητα παντού <clears throat> στις χώρες της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης να υπάρξει συμφωνία για ένα ελάχιστο επίπεδο αμοιβών, για μια, ένα ελάχιστο κοινωνικό μισθό. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο για τα θέματα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε για τα ελάχιστα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων στην Οικονομική Νομισματική Ένωση. Για μένα αυτό είναι κάτι το θεμελιώδες να υπάρχει ένας ελάχιστος νο, επίσημος κοινωνικός μισθός σε όλα τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ. Γιατί αλλιώς θα χάσουμε την υποστήριξη όλων των, των εργατικών στρωμάτων, αν θέλετε να το πω λιγάκι, <clears throat> με αριστερή μαρξιστική φρασιολογία. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε και ποια είναι η έννοια, το περιεχόμενο της αλληλεγγύης που περιλαμβάνεται και στην έκθεση Φαν Ρομπάι. Πρέπει να συμφωνήσουμε όχι μόνο για την αρχή, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί αυτή η αλληλεγγύη. Και να ξέρουμε ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές ενός συστήματος εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων. Δεν μπορούμε να έχουμε την ε, τραπεζική εποπτεία, την ενιαία τραπεζική εποπτεία για την οποία έχουμε κάνει τεράστιες προόδους και έχουμε και κάποιες πρώτες σκέψεις για το μηχανισμό επίλυσης τραπεζών και το Ταμείο Εγγύησης των, ε, των ε, τραπεζικών κατεθέσεων στην περίπτωση της Ελλάδος και η Σάρου θα με ρωτούσε ίσως και για την Κύπρο καταφέραμε χάρη στην ε, αποφασιστικότητα της ε, ελληνικής κυβέρνησης και χάρη στην ε, προσπάθεια και του ελληνικού λαού που επλήγηκε τα μάλα στα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα από την εφαρμογή αυτού του συστήματος του, των ενεργειών για την σταθεροποίηση και την εξυγίανση των οικονομικών. Μιλάμε πάρα πολλέ φορέ για το 2 το 6 δεν μιλάμε πάντα για τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λαοί. Uh, um, Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε λίγο πίσω στον χρόνο. Θα μας βοηθήσουν όμως οι ευρωβουλευτές εδώ. Εκτός αν είμαστε εδώ ακόμα μέχρι τις 2. Θα δούμε. Πρώτα απ' όλα, εκ του ΕΛΚ, ο Ζαν Πολ Γκοζές. Ζαν Πολ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, δεν θα μιλήσω πολύ χρόνο, οπότε θα κερδίσουμε από την καθυστέρηση αυτή. Εκ μέρου των συναδέρφων από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θέλω να σου πω ότι ήταν μεγάλη χαρά η συνεργασία μας. Δεν είναι θέμα διάθεσης νοσταλγικής, απλώς πιστεύω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό, θεμητό, τώρα που θα δώσετε την προεδρία της Κιτάλη σε κάποιον άλλον που δεν είναι τόσο γνωστός, να σας πούμε ότι έχουμε εκτιμήσει πάρα πολύ τη συνεργασία μαζί σας, σε όλες τις συναντήσεις μας και όλα όσα έχετε κάνει στο Eurogroup. Μάλιστα επιτρέψτε μου να σας πω, Ζαν ότι πριν αναφέρθηκα στους σοφούς. Εγώ νομίζω ότι ναι. Το όνομα του σοφού νομίζω ότι μπορείς κάλλιστα να το έχεις. Γιατί είσαι ένας σοφός μη κομφορμιστής, κάτι το οποίο επέτρεψε στις διάφορες συναντήσεις να είναι τόσο ζωντανές και να μπορέσουν όλοι έτσι να καταλάβουν καλύτερα ποιος ακριβώς είναι ο προβληματισμός και προς ποια κατεύθυνση θέλεις να πάμε. Τώρα για να κερδίσουμε χρόνο. Μην πω τώρα στην Ευρωζώνη και την Ευρώπη. Να σου πω όμως το εξή ότι στη Γαλλία έχουμε το εξή φαινόμενο. Ακούμε την κυρία Μέρκελ, η οποία μας, επιτρέ... μας ε, υπόσχεται δύσκολα χρόνια ακόμα προκειμένου να βγούμε από την κρίση ενώ από την άλλη μεριά ακούμε τον κύριο Όλαντ να μας λέει ότι τελείωσε η κρίση, ότι έχουν περάσει τα πιο δύσκολα και θα φανεί αυτό στα τέλη του 2013. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε μια διφωνία, ακούμε δύο διαφορετικά πράγματα και θα ήταν ενδιαφέρον εσύ να μας πεις μια που είπαμε ότι δεν είσαι κοφορμιστής, ποια άποψη έχεις γι' αυτό. Τρία λεπτά σας μένουν. Δεν χρειάζομαι τρία λεπτά γιατί κατάλαβα τι υπονοεί ο κύριος Γκοζές με την ερώτησή του. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι ανάμεσα στην κυρία Μέρκελ και τον κύριο Λάουντερ υπάρχουν όλες αυτές οι αποχρώσεις, οι μουσικές στις οποίες εσύ αναφέρθηκες όταν μίλησες για διφωνία. Οι σχέσεις Γαλλίας-Γερμανίας ε, ποτέ δεν εντυπωσίαζαν από την ποιότητά τους τους ε, μουσικόφιλους. Η συνεννόηση ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις είναι ικανοποιητική. Θα μπορούσαν να ήταν καλύτερη. Αλλά εδώ και δεκαετίες ισχύει αυτό. Εκτός όταν ε, κάποιοι αποφάσισαν να συντονίσουν την ορχήστρα και το έκαναν με νοσταλγική διάθεση. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι οι επόμενες χρονιές θα είναι δύσκολες. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει έτσι με ωραία λόγια να καλύπτουμε την ανάλυση μας. Πιστεύω ότι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε παραμένουν. Είναι σοβαρά προβλήματα. Η λύση τους απαιτεί μεγάλη δόση θάρρους, πολιτικού θάρρους. Όμως δεν θα ήθελα από την άλλη μεριά να στηρίξω τις φωνές εκείνες Ότμαρ μιλάει. Όταν μιλάς σε παρακαλώ να μιλάς πιο, πιο χαμηλά. Δεν κατάλαβες έτσι γιατί δεν ε, ακούγησα πολύ δυνατά. Εκτός μικροφώνου παρέμβαση. Ναι. Αν αλλάζει τώρα η παρτιτούρα βέβαια, αλλάζει και η μουσική. Έλεγα λοιπόν ότι ανεξάρτητα από όλες αυτές τις ε, μουσικές συζητήσεις, θα ήθελα να σας πω ότι εγώ πιστεύω ότι εξακολουθούν να είναι δύσκολοι οι καιροί και ότι δεν θα πρέπει να δώσουμε την εντύπωση στην κοινή γνώμη των χωρών μας, στα Εθνικά Κοινοβούλια, ότι ε, τα... οι δύσκολοι καιροί έχουν τελειώσει. Μπορεί τα πιο δύσκολα να βρίσκονται πίσω μας, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε δυσκολίες και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Ωραία, λέει. Η Πρόεδρος, αυτή ήταν η σύντομη ερώτηση, πήρε πέντε λεφτά. Ε, ο Ότμαν φταίει. Ότμαν φταίει, λέει και η Πρόεδρος. Ελίζα. Κύριε Πρόεδρο, εξ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, <clears throat> θα ήθελα και εγώ να σας πω ότι ακόμα και όταν διαφωνούσαμε, ποτέ δεν αμφισβήτησα την πείρα σας και την ικανότητά σας. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι ήσασταν επικεφαλής της ζώνης του ευρώ σε μια τόσο δύσκολη εποχή. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα, <clears throat> το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά εγώ θα σταθώ τώρα σε κάποιο άλλο ζήτημα, που είναι το θέμα των αρμοδιοτήτων του, της Ευρωομάδος και του Πρόεδρου αυτής της ομάδος έναντι των χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα δημοσιονομικής σταθερότητας. Το ερώτημά μου έχει να κάνει με τα έσοδα, <clears throat> με τις συνταγές οι οποίες προτείνονται. Είναι πολλές χώρες, δεν είναι λίγες, οι οποίες ακολούθησαν κατά γράμμα τις επιταγές για την... Ε, για την ε, έχετε πρόβλημα με τη μετάφραση, για την σταθεροποίηση των δημοσιονομικών τους. Δεν είναι πρόβλημα η ίδια η σταθεροποίηση το πρόβλημα το οποίο εγώ θέλω να θέσω είναι το πρόβλημα του ρυθμού αυτή τη δημοσιονομική σταθεροποίηση και των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει. Γιατί πολλέ χώρε ακολούθησαν κατά γράμμα αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί, ελπίζοντα ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή μια μείωση τη ανεργία και αύξηση τη οικονομική μεγέθυνση και είδανε τελικά ότι έχουν μια ύφεση 3-4% και συγχρόνως ανεβαίνει η ανεργία και αυτό σημαίνει και μεγάλα και σοβαρά προβλήματα κοινωνικού χαρακτήρα. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να ξαναδούμε αυτές τις συνταγές, αν μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε τον ρυθμό ε, αναπροσαρμογής των οικονομιών και εδραίωσης των δημοσιονομικών. Κυρία Πρόεδρε, θα έλεγα στην Ελίζα που μαζί προχωράμε εδώ και τόσα χρόνια ότι και εγώ έχω πολλά ερωτηματικά για το ρυθμό με τον οποίο προχωράνε αυτά τα προγράμματα στις διάφορες χώρες. Γενικά, όχι εσείς, αλλά σίγουρα διάφορες κυβερνήσεις βλέπουν τεράστια ανεργία στις χώρες τους, η οποία πραγματικά είναι τεράστιο βάρος για μας, πάνω από 11% στην Ευρωζώνη. Ενώ υποσχεθήκαμε στους Ευρωπαίους ότι τα πλεονεκτήματα μας είναι μοναδικά και έτσι θα υπάρχουν κοινωνικές ισορροπίες και δικαιοσύνη για τους εργαζόμενους. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι οι άνεργοι αυξάνονται, ότι οι άνεργοι είναι εντάξει δεν θα έλεγα ακριβώ ο κανόνας, αλλά πάση περιπτώσει όχι και η εξαίρεση. Οπότε θα έπρεπε σε όλε μα τις χώρες και σε ολόκληρη την Ευρώπη να έχουμε πιο δραστήριες πολιτικές σε σχέση με την αγορά απασχόληση. Δεύτερον, εγώ συμφωνώ με τη σχολή εκείνη, η οποία είναι βέβαια μειοψηφία στην Ευρωζώνη, η οποία θα ήθελε οι χώρες που προχωράνε σε διαρθρωτικές προσαρμογές, όπως η Πορτογαλία, αλλά είναι και η Ελλάδα βέβαια στην ίδια κατηγορία και η Ιρλανδία και η Ισπανία και η Ιταλία, αλλά πάση περιπτώσει μιλάω πιο συγκεκριμένα για τα μνημόνια, οπότε Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία κυρίως. Θα έπρεπε λοιπόν εκεί να έχουμε ένα σύστημα, και δεν το λέω αυτό με πατερναλιστική διάθεση, ε, αντιστάθμισης, έτσι αποζημίωσης, επιβράβευσης κατά κάποιο τρόπο στις χώρες εκείνες οι οποίες κάνουν την προσπάθεια. Το έχω προτείνει πολλές φορές, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Πορτογαλίας, να ξαναδούμε τον μηχανισμό ε, οικονομικής προσαρμογής και τη δημοσιονομική προσαρμογή. 4 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα, κυρία Πρόεδρε. Ε, ξεκίνησε λοιπόν ανταγωνισμό τώρα. Για να δούμε τώρα πώς θα συνεχίσει το, η επόμενη ομάδα. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν είσαστε σοφός. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι είσαστε ένας πεπισμένος Ευρωπαίος. Έχετε τονίσει και έχετε κάνει ορατό το ότι η Ευρώπη έχει πράγματι μια καρδιά και εμείς ως φιλελεύθεροι σας υπεστηρίζουμε απόλυτα σε αυτό. Δύο ερωτήματα το θέμα της εσωτερικής αγοράς και της ε, παγκοσμιοποίησης. Έχουμε κάνει μια πρόοδο στα θέματα αυτά. Υπάρχουν πολλά κράματα, κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρούν ότι είναι επαρκής Θεωρούν ότι είναι επαρκή η ολοκλήρωση τη εσωτερική αγορά. Για πολλέ χώρε τη Ευρωζώνη δεν είναι αυτό έτσι. Βλέπετε να υπάρχει ένα κίνδυνο, να υπάρξει μια κατά κάποιο τρόπο μορφή απο, αποσύνδεσης της Ευρωζώνης και τη υπόλοιπη ε, Ευρώπη επίση. Τους τελευταίους μήνες έχουν ξεκινήσει πολλά σημαντικά σχέδια, αλλά συνήθως χωρίς τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου έχουν χρησιμοποιήσει μια καθαρά διακρατική μέθοδο. Για μας αυτό δεν είναι το πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας. Πώς τα κρίνετε όλα αυτά τα γεγονότα. <clears throat> Για τα δύο αυτά ερωτήματα τα οποία έχει θέσει ο Βόλφ. Εγώ πάντα έχω προσπαθήσει να μην δημιουργήσω χάσμα μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ και των χωρών που είναι έξω από τη ζώνη του ευρώ. Έτσι, όπως την διατυπώνεται αυτή την ερώτηση, ξέρουμε ότι υπάρχουν, ότι υπάρχουν κάποιες δυνάμεις οι οποίες έχουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν δεχθεί να μπουν στη ζώνη του ευρώ και υπάρχουν χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία που παραμένουν στα πλαίσια του opt-out. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις χώρες εκτός της ζώνης ευρώ με διαφορετικό τρόπο. Είναι άλλη η Δανία, άλλο το Ηνωμένο Βασίλειο, άλλη η Τσεχική Δημοκρατία. Γι' αυτό υποστηρίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτήν την αρχιτεκτονική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δύο χώρε οι οποίε δεν θέλουν με κανένα τρόπο να είναι τμήματα τη Ευρωζώνη. Υπάρχουν πολλέ άλλε οι οποίε θέλουν να γίνουν καιρό μέλη τη Ευρωζώνη. Δεν μπορούμε να έχουμε μια αδιαφοροποίητη λοιπόν αντιμετώπιση για όλε αυτέ τι χώρε. Και εγώ συμφωνώ μαζί σα ότι πρέπει να φτιάξουμε νέα τύχη μέσα στην Ευρώπη στην αρχή του 21ου αιώνα. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι το κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι ένας ε, πυρήνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ακολουθήσει πλήρως την ενωσιακή μέθοδο και όχι να παραμείνει στα πλαίσια της ε, διακρατικής μεθόδου. Αυτό δεν οδηγεί μονάχα σε ένα θεσμικό χάος η διακρατική μέθοδος, αλλά οδηγεί και σε μια σύγχυση στην συνείδηση των πολιτών. Εγώ έχω φτάσει στο σημείο αυτό που έχω αναφέρει αυτό, αυτό που είπε ο Κομφούκιος ότι όταν χάνουμε τις λέξεις τότε ακολουθεί το χάος. Ο Κομφούκιος το είπε, όχι εγώ. Για να σας ε, αναφέρω κάποιον ο οποίος είναι πράγματι σοφός. Αν θέλεις να ε, επανέλθεις, έχεις, υπάρχει χρόνος. Επειδή είσαστε και μου ζήτησε μια, μου ζήτησε μια γείτονά μου να θέσω το θέμα τη ε, ισότητα των φύλων. Γιατί όπω ξέρετε υπάρχει το θέμα ότι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν υπάρχει καμία γυναίκα στο Διοικητικό Σύμβουλο. Πώ τα βλέπετε τα θέματα αυτά, ιδίω με τα νέα εποπτικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ κατανοώ την, ε, τις ανησυχίες της Επιτροπής Γυναικών και τη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν σαφείς. Έχω απόλυτη κατανόηση για το γεγονός αυτό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει με μεγάλη δυσκολία δεχτεί την εκλογή μελών που δεν ήταν ε, γυναίκες. Έχουμε συζητήσει για το θέμα αυτό επανειλημμένα. Πρέπει να πω ότι και πριν από τα πρόσφατα ε, συμβάντα τα οποία σε έβαλαν σε αμήχανη θέση, είχες ε, εκφράσει συμφωνία με την απόψή μας. Ε, θυμάμαι όταν είπες ότι ίσως ε, ίσως ε, θα πρέπει να απορρίψουμε κάποιον και εσύ είπες μακάρι. Ωραία. Λοιπόν, ECR. Να προσθέσω δύο λόγια. Μία, μία φράση μόνο. Εγώ απολύτως θέλω να υπάρχουν ε, γυναίκες ε, εκπρόσωποι όχι μονάχα στο, ε, εδώ αλλά και σε όλους τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μακάρι να είναι, αλλά θα είναι και θα είναι Γαλλίδα. Right. ναι, ναι, κάτι κατάλαβες, κάτι κατάλαβες εσύ, κάτι ξέρεις. Κύριε Γιούγκερ, την θέση αυτή που είχατε για 8 χρόνια θα την εγκαταλείψετε εν καιρό. 8 χρόνια για ένα πολιτικό είναι αιωνιότητα. Ίσως όχι στο Λουξεμβούργο, αλλά στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι. <clears throat> Ποιο είναι το πιο σημαντικό δίδαγμα το οποίο έχετε αποκομίσει ως επικεφαλής της Ευρώπη. Τι είναι αυτό το οποίο έχετε μάθει αυτά τα τελευταία 8 χρόνια. Δεύτερον, ποιε θα πρέπει να είναι οι προσωπικές ικανότητες και ιδιότητες που θα έχει ο διάδοχός σας ποια είναι η άποψή σας για τον ε, προτινόμενο διάδοχό σας και ποια διδάγματα θα του μεταφέρετε. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για το έργο σας και να σας ευχαριστήσω καλή τύχη στο όμορφο Λουξεβούρ. Die Deutschen, wenn sie denken, hört nicht zu. Ε, <laughs> οι, Γερμανοί όταν δεν τους ακούει κανείς κάνουν κάποια σχόλια για το μέγεθος της χώρας μου. <laughs> Εμείς δεν είμαστε ούτε Γερμανία ούτε Ηνωμένο Βασίλειο και θα πρέπει να ζήσουμε μέσα στα δικά μας μέτρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αφήνουμε να μας παρασύρουν οι συγκινήσεις, η συναισθηματική προσέγγιση και γι' αυτό καταφέρουμε να επιβιώσουμε όλα αυτά τα χρόνια για τον ναι, διάδοχό μου. Δεν έχω να δώσω κάποια επίσημη δημόσια συμβουλή να του δώσω. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα ευτυχές και επιδέξιο. Στην, ε, σε προσωπικό επίπεδο θα μπορούσα να του πω ότι πιστεύω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα πρέπον και αρμόζον να αναφέρω προσωπικές, ε, επισήμ, επισήμως προσωπικές μου απόψεις αυτού του είδους. Θα πρέπει μόνος του να αποφασίσει τι είναι το καλύτερο. Δεν, είμαι, δεν, έχω πια τέτοια, δεν έχω ακόμα τέτοια απόσταση που να μπορώ να σας ε, παρουσιάσω ένα απολογισμό για τα τελευταία 7 χρόνια που ήμουν επικεφαλής της Ευρωομάδος. Γιατί αν ε, τα κάνω ε, αυτή τη στιγμή και αυτοσχέδια μπορεί να βγουν μονάχα τα αρνητικά στοιχεία. Γιατί στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή έχω όλα τα στοιχεία τα οποία <clears throat> δεν πήγανε καλά. Όλες τις αποτυχίες, όλες τις αποφάσεις οι οποίες δεν ήταν επιτυχείς, όλα τα στοιχεία καθυστέρησης είτε ε, εν γνώση μας είτε μη εν γνώση μας αναγκαστήκαμε να δεχτούμε που θα μπορούσε να είχαν βοηθήσει μια ταχύτερη λύση της κρίσης. Ίσως τα πράγματα τα οποία είναι θετικά θα έρθουν αν σκεφτεί κανείς λίγο περισσότερο χρονικό διάστημα. Και έχω και μια σκέψη η οποία από τότε που ξεκίνησα να είμαι πολιτικός σε ευρωπαϊκό επίπεδο πριν από δεκαετίες, ότι θα πρέπει να μην υποτιμούμε την πολυπλοκότητα της Ευρώπης. Ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε να ακούμε και τις απόψεις και να λαμβάνουμε υπόψη τις ευαισθησίες και των άλλων. Όταν έρχεται κανείς από το μικρό Λουξεμβούργο είναι καταδικασμένος να ακούει τις απόψεις των άλλων. Και ξέρω ότι οι γείτονέ μας δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το Λουξεμβούργο, μπορούν ε, να μας κοροϊδεύουν ε, ή να κάνουν αστεία για μας. Αυτό, επομένως, μας κάνει να σκεφτόμαστε με ένα διαφορετικό τρόπο. Η γνώση αυτή πιστεύω ότι είναι πολύ πολύτιμη για να μπορεί κανείς να καταλάβει την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα είναι και συμβουλή μου. Αν θέλετε, τώρα που το σκέφτηκα θα μπορούσε να είναι αυτή η συμβουλή που θα δώσω στον ε, ε, διάδοχό μου. Θα πρέπει να δέχεται και να αγαπάει τις απόψεις των άλλων. Επίσης, ε, είπατε ότι πρέπει το χρόνο του και αυτό είναι ενδιαφέρον. Θα το δούμε ως Και από μας ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα λόγια που έχετε αναφέρει όχι μόνο εδώ αλλά και σε, άλλους, σε άλλα βήματα και για τη σαφή δέσμευση που έχετε αναλάβει και φέρει σε πέρας για να υπάρχει μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή δομή και ευρωπαϊκή ιδέα. Και επίσης για όλα αυτά που είπατε για τις κοινωνικές αστοχίες που ήταν τμήμα όλου αυτού του εγχειρήματος οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Τώρα, μετά από τους επένους θέλω να σας πω και κάτι το οποίο ίσως είναι πιο επικριτικό. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μεγάλο ενδιαφέρον να υπάρξουν από το Συμβούλιο και την Κομισιόν οι κατευθυντήρες γραμμές για δύο χώρες, μία από τις οποίες είναι η Αυστρία και η άλλη είναι το μεγάλο δουκάτο του Λουξεμβούργου και να μπορέσει να ε, αντιμετωπιστεί επίσης το θέμα της ε, ανταλλαγή ανταλλαγής στοιχείων με τις Ηνωμένε Πολιτείε όταν υπάρχει λοιπόν παράδοση στοιχείων σε μια τρίτη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζω ότι θα μπορέσει να επιληθεί το θέμα αυτό. Έχω ένα παρεπεραιτέρω ερώτημα. Αν θέλετε ένα, ένα δώρο αποχώρησης, μήπως θα μπορούσατε με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσετε ότι η οδηγία που ανέφερα προηγουμένως θα γίνει δεκτή, θα γίνει δεκτή και θα εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες και επίσης να αντιμετωπιστεί το θέμα των ποσών που χάνονται σε φορολογικούς παρα, παραδείσους. Εγώ χαίρομαι για το πρώτο τμήμα της παρέμβασής σας, για τους επένους σας. Και εγώ θέλω να σας ε, συγχαρώ για όλα αυτά. Ίσως έχω κάποιες διαφορετικές απόψεις σε ορισμένα σημεία. Ήσασταν πάντα ιδιαίτερα αυρόφρον. <laughs> Δεν χρειάζεται λοιπόν να ζητήσετε συγγνώμη για αυτό, για το δεύτερο σημείο. Το, τη δεύτερο, το δεύτερο τμήμα του για την ε, οδηγία αυτή για τα επιτόκια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει. Είναι περισσότερο βέβαια θέμα του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ, όχι της ε, Ευρωομάδος. Είδα ότι στο γερμανικό τύπο αναφερθήκαν πάρα πολλά θέματα για τα αυτά και θεωρήθηκε ότι σε αυτό υπήρξαν και κάποιες δηλώσεις του αρμοδίου επιτρόπου σε σχέση με μένα που δεν ήταν ιδιαίτερα κολακευτικές. Παρακαλώ. Όχι, όχι, μην, ε, μην χρησιμοποιείτε αποδοκιμαστικές εκφράσεις. Το Λουξεμβούργο λοιπόν πάντα σας εκπλήσει. Υπάρχει αυτή η οδηγία για τα επιτόκια μόνο γιατί η Προεδρία του Λουξεμβούργου είχε στο παρελθόν ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία της οδηγίας με στόχο να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή. Γιατί το Λουξεμβούργο είχε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, γιατί είχε χάσει με αυτή τη διαδικασία πολλά φορολογικά έσοδα. Εγώ όταν ήμουνα ε, Υπουργό Οικονομικών ήξερα καλύτερα το σύστημα το φορολογικό των κάτω χωρών από ότι το λουξεμβουργικό και έβλεπα ότι υπήρχαν και από άλλες χώρες για προτάσεις για το τι έπρεπε να κάνει το Λουξεμβούργο για την πολιτική αυτή. <laughs> οι μεγάλες χώρες οι οποίες είναι ε, ένοχες κατά κάποιο τρόπο μέσα εισαγωγικά στα φορολογικά θέματα είναι πολύ πιο μικρές από τις μεγάλες χώρες, οι οποίες είναι μικρότεροι φταίχτες στα θέματα αυτά. Τα θέματα του φόρου ΦΠΑ, του φόρου ε, κατανάλωσης, του φόρου της φορολόγησης των τόκων, όλα αυτά τα θέματα τα αντιμετώπισε το Λουξεμβούργο. Και γι' αυτό εκπλήσωμαι όταν λένε «Α, το Λουξεμβούργο είναι ένα μέρος όπου κυκλοφορεί μαύρο χρήμα, γίνεται ξέπλυμα χρήματος, είναι φορολογικό παράδεισος». Αυτά δεν ήταν ακριβώς αυτά που κάναμε. Πολλοί μας τα λένε αυτά γιατί ακριβώς εμείς πολλές φορές ξέρουμε περισσότερο για αυτούς από ότι αυτοί για τον εαυτό τους. Για την οδηγία, για τα επιτόκια συγκεκριμένα το Λουξεμβούργο θα σας εκπλήξει και θα σας εκπλήξει θετικά το λέω. Δεν έχουμε χρόνο να ε, ξαναπάρουμε τη συζήτηση αυτή. Η Γκούε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ εξ ονόματο τη ομάδα μου θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας ευχαριστήσω και για την παρουσία σας εδώ σήμερα και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό σε ένα σημείο το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως και ήταν από τα θέματα συζήτησης στην επαφή μαζί σας. Θέλω να μιλήσω και για τα προβλήματα προσαρμογής γιατί εμείς έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση για τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται συγκεκριμένα στη δική μας χώρα, στην Πορτογαλία το έγγραφο το οποίο έχει έρθει εδώ είναι σαφές ότι δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί οι στόχοι οι οποίοι έχουν αναφερθεί για την Πορτογαλία για την αντιμετώπιση της ε, έλλειψης φορολογικών εσόδων και παρόλα αυτά, παρά το γεγονός ότι είναι σαφέ ότι υπάρχουν προβλήματα, η απάντηση που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι. Γνωρίζετε την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που αναφέρει ότι οι μέθοδοι που προτείνονται για την Πορτογαλία οδηγούν σε περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, σε περαιτέρω απολύσεις, σε περικοπές στην υγεία και την εκπαίδευση. Όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα τα οποία περιλαμβάνονται στο, στο πρόγραμμα σταθεροποίησης οδηγούν σε, σε θέσεις οι οποίες ουσιαστικά ανασκευάζονται από οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά ούτως ή άλλως είναι φορείς οι οποίοι δεν έχουν νομο, δημοκρατική νομιμοποίηση. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω το θέμα αυτό μετά από τα χρόνια που ήσασταν επικεφαλής της Ευρωομάδας. Βλέπετε αυτή τη στιγμή να υπάρχει η καταστροφή του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη. που ησασταν επικεφαλη της γίνεται αυτή η καταστροφή από θεσμούς που δεν έχουν δημοκρατικό έλεγχο. Γι' αυτό έχουμε φτιάξει το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Εκεί μας οδηγεί το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σας θέση και πώς απαντάτε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. I'm invited to be short. Λοιπόν, συμμερίζομαι τις ανησυχίες, σας, τις ανησυχίες σας, αλλά όχι τα συμπεράσματά σας όλα. Αναρωτιέμαι και εγώ όσον αφορά την δημοκρατική ποιότητα των ε, φορέων ε, του Συμβουλίου που μας προτείνουν να πάρουμε κάποια μέτρα. Το ίδιο ισχύει και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, και για την Κεντρική Τράπεζα και το ίδιο ισχύει και για την Κομισιόν. Και για τον ΟΣΑ επίσης, αλλά δεν είναι το τέταρτο μέλος της Τρόικα. Έστω και αν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι ε, ο ΣΑ έχει ήδη βάλει το πόδι του μέσα οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Eurogroup. Εμείς δεν μπαίνουμε ποτέ στις λεπτομέρειες των μέτρων που αναλαμβάνουν ε, τα, ε, χώρε, οι χώρες μέλη της ε, Ευρωζώνης ή οι άλλες χώρες. Πάντα έλεγα ότι η μέθοδος αυτή δεν είναι η μεθοδος αυτη δεν ειναι βελτιστη Θα έπρεπε να έχουμε την δυνατότητα εν λεπτομερία να μελετούμε τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και θεωρώ ότι κάποια από τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν κυρίως στην Ελλάδα είναι μέτρα τα οποία τελικά, ε, ε, τελικά έχουν κακά αποτελέσματα στους λιγότερο ε, κατέχοντες και όχι το αντίθετο. Και αυτού του είδους τα μέτρα δεν είναι σωστά, τα καταδικάζω. Απ' την άλλη πλευρά, οι αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης να μεταφέρουν, της μεταφοράς κεφαλαίων προς το Λουξεμβούργο, προς τη Γερμανία, προς την την Φραγκφούρτη, προς, ε, ε, προς το Λονδίνο, ε, θέμα το οποίο φαίνεται ότι οι Γερμανοί το παραβλέπουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη και αυτές οι αρχές, οι απανταχού της Ευρώπης, θα πρέπει με τον καλύτερο τρόπο να συνενέσουν και να βοηθήσουν να συνδράμουν την ελληνική κυβέρνηση, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η μη πατριωτική συμπεριφορά των εκατομμυριούχων και πολυεκατομμυριούχων Ελλήνων ή τουλάχιστον ορισμένων μεταξύ αυτών. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια ε, τα μέτρα τα οποία αναλαμβάνονται. Πολλές φορές έχω πει ότι και εγώ ο ίδιος θα είχα προτείνει την ε, μείωση του ελάχιστου μισθού ε, στην Ελλάδα. Εγώ δεν ήμουνα καθόλου σύμφωνος όταν συζητήθηκε το θέμα αυτό στο Eurogroup, αλλά δεν μπορούσα να κάνω και κάτι. Ε, θα πρέπει να γίνουν πιο δημοκρατικές και πιο συμφιλιωτικές ε, οι αποφάσεις μας επί των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν. Ε, κοιτάξτε, εδώ είμαι για τελευταία φορά, επομένως ίσως μπορώ να ξεπεράσω και λίγο το χρόνο μου. Πρόεδρος. Το, πρόβλημά μου είναι ότι ήδη έχουμε ξεπεράσει κατά 25 λεπτά το πρόγραμμά μας και θα μείνουν μερικοί απογοητευμένοι. Ε, αλήθεια είναι ότι αργήσαμε να ξεκινήσουμε γιατί μέχρι να πούμε χρόνια πολλά ο ένας τον άλλον ε, μας πήρε πολύ χρόνο. Ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε που για τελευταία φορά έρχεστε εδώ. Κατά τη διάρκεια της ευρωκρίσης ε, η ευρωζώνη ε, κατά περιπτώσεις ε, δεν είχε κοινή πολιτική. Ο Βορράς και ο Νότος συχνά διαιρέθηκαν όσον αφορά την είχαν διαφορετική άποψη σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης. Βεβαίως είναι εμπειρασμένη η ευθύνη των, και του χρέους ακόμα. Βλέποντας τα τελευταία χρόνια της θητείας πώς βλέπετε αυτό, αυτή την απόκληση Πώς βλέπετε ε, τα πράγματα για το μέλλον, ποιες προβλέπετε δηλαδή να είναι οι εξελίξεις απάντηση. Είναι γεγονό ότι ξεκίνησε λίγο αργά, ε, μάλλον με κάποια καθυστέρηση η συνεδρίαση, ε, γιατί είχαμε ε, πολλά, πολλά, πολλές χαιρετούρες στην αρχή. Όταν έρχεται ο πρόεδρος Ολάντε και όταν έρχεται και η καγκελάριος Μέρκελ, καθυστερούμε γιατί μπλοκάρονται όλοι στην είσοδο για να γίνει ο έλεγχος. Εγώ δεν έχω, έρχομαι μόνος μου και μόνο χαιρετάω όλο τον κόσμο. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και χώρες του Νότου. Ε, αυτοί που κάνουν αυτό το, το διαχωρισμό είναι αυτοί του Βορρά και αυτοί του Νότου. Υπάρχουν όμως κάποια αντικειμενικά μέτρα και κάποιες αντικειμενικές βάσεις για την ε, συζήτηση που πρέπει να γίνει. Πιστεύω ότι και ο Βορράς και ο Νότος και η Ανατολή και η Δύση πρέπει να κινηθούν ομού αυτοί του Βορρά ή αυτοί από το Βορρά που θεωρούν ότι είναι πολύ πιο ενάρετοι από αυτούς του Νότου, θα πρέπει να δουν λίγο τα του οίκου τους, να δουν λίγο πώς εξελίχθηκαν τα νούμερα τα τελευταία χρόνια και θα ανακαλύψουν ότι δεν είναι και τόσο ενάρετοι δά όσο νομίζουν. Και αυτοί του Νότου, αυτοί που θέλουν να μπαίνουν και να μένουν σε αυτή την κατηγορία, κατέβαλαν πολλές προσπάθειες έτσι ώστε να μπουν ε, στην Ευρωζώνη. Ας θυμηθούμε την κατάσταση της Πορτογαλίας, της Ιταλίας ε, κάποια χρόνια ε, πριν ήταν τότε πολύ πίσω από άλλες χώρες και έκαναν τρομακτικές προσπάθειες, κατέβαλαν μεγάλες ειλικρινά προσπάθειες έτσι ώστε να φτάσουν στο σημείο να ε, μπουν στο Eurogroup. Γι' αυτό δεν θέλω αυτούς τους διαχωρισμούς ε, και επιμένω και επαναλαμβάνω δεν είναι πιο ενάρετες οι χώρες του ε, Βορρά και οι χώρες του Νότου δεν είναι πιο αμαρτωλές από αυτές του Βορρά. Ευχαριστώ συμφωνώ και εγώ και χαίρομαι που μπορώ να μεταφέρω αυτά τα μηνύματα στην ε, Φιλανδία. Ναι, ε, η Φιλανδία νομίζω ότι θα ήταν ένας καλός αποδέκτης αυτού του μηνύματος. E Είχατε πει στην πρώτη σας ε, απάντηση ότι έστω και αν κάποια πράγματα έχουν ήδη δύσκολα, έχουν ξεπεραστεί, Ποιε είναι οι δύσκολες αποφάσεις που ακόμα απομένουν. Απάντηση. Δεν νομίζω ότι, ότι μπορούμε να μιλήσουμε για ε, επιπλέον ε, προβλήματα ή να εξειδικεύσουμε το θέμα στις, ε, στα συστήματα ασφάλισης κτλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα ανάπτυξης και το δυναμικό ανάπτυξης της κάθε χώρας θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι θα αντιμετωπίσουμε όλοι σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά μας συστήματα και τα συστήματα πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης συγγνώμη, για τα, ε, τις επόμενες δεκαετίες ε, τα ε, συστήματα τα οποία εφαρμόζονται από δημοσιονομικής πλευράς δεν είναι εύκολα επιβιώσιμα, κατά κάποιο τρόπο η επιβίωσή τους δηλαδή είναι αμφίβολη και το δεύτερο σημείο που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά πιστεύω ότι θα πρέπει να ανακαλύψουμε μια βιομηχανική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν έχουμε κάτι τέτοιο, δεν έχουμε βιομηχανική πολιτική. Αυτό συνδέεται, όχι αποκλειστικά βέβαια, ε, ε, στον τομέα της χαλιβουργίας. Έχουμε χαλιβουργική παραγωγή ε, η οποία ε, βασίζεται, ε, αν τα πράγματα πάνε καλά, σε 12 εκατομμύρια τόνους. Εάν οι μειώσεις οι οποίες επιβάλλονται ε, ε, με, τις, ε, με τους περιορισμούς που επιβάλλουν φτάσουμε στους 140, τότε δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει αποδεκτό χωρίς πολιτικές έτσι, αναταράξεις. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο και όλο το θέμα της εργασίας και της αντιμετώπισης της, αλλά αυτό είναι πολύ πιο περίπλοκο και δεν είναι τη στιγμή. Λοιπόν, Μάρτιν, ε, θα πρέπει τέσσερα λεπτά το πολύ να κρατήσει η ανταλλαγή αυτή, γιατί αλλιώς θα μείνουν πολύ ε, απογοητευμένοι. Εγώ δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω τα πέντε λεπτά. Γνωριζόμαστε από το 1997. Είχαμε συζητήσει τότε με τον τότε καγκελάριο Κλιμ της Αυστρίας για τα θέματα της παγκοσμιοποίησης που είχε πει ότι η παγκοσμιοποίηση δίνει τεράστιες ευκαιρίες αλλά αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά θα οδηγήσει σε ανισότητες στην ανάπτυξη και σε δημοκρατικά ελλείμματα. Και είχε τονίσει από τότε ήδη τη σημασία της, του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Δυστυχώς δεν. <laughs> Δυστυχώς είχε στη λάθος δουλειά είσαι ένας χαρισματικός εμπειρογνώμων και ικανός να πείθεις τους άλλους όσο υπάρχουν πολύ λίγοι και είσαι και ένας μεγάλος ευρωπαϊστής. Το λάθος ήταν ότι υπήρχαν πολύ λίγοι Λουξεμβούργοι σαν και σένα οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θα προτιμούσαν να έχουν εσένα ως πρόεδρο της Κομισιόν το 1999, το 2004, το 2009. θα έπρεπε να φανταστεί κανείς πώς θα είχε εξελιχθεί η Ευρώπη με τον jean Κλοντ Juncker και όχι με τον τωρινό πρόεδρο, με τους τωρινούς πρόεδρους. Εσύ είχε πάντα τις ιδέες και τα οράματα αυτά. Θα μπορούσε να είχε δοθεί μια όθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έκανε τους Αμερικανούς να μας Και εδώ το πρόβλημα είναι ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αυτό είχε τεράστιες συνέπειες. Γιατί είναι πολύ λίγοι αυτοί που είναι σαν και σένα και οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν αυτό το οποίο έκανες εσύ. Να αποφύγουν να υπάρξει μια διάσπαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διατηρήσουν το ενωσιακό σχήμα έναντι του διακρατικού ε, συστήματος λήψης αποφάσεων. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι αν ήταν επικεφαλής ο Jean-Claude Juncker, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα είχαμε αντιμετωπίσει μια τόσο μεγάλη κρίση. <clears throat> δεν θα είχαμε καθυστερήσει τόσο πολύ ε, για την εμβάθυνση της Ευρώπης, δεν θα είχε υπάρξει μια τόσο μεγάλη κα, ε, καθυστέρηση. Δεν θα είχαμε λοιπόν όλη αυτή την ασάφεια σε σχέση με πολιτικούς στόχους. Θα είχαμε πει με αυτές τις προϋποθέσεις θα έρθουν όλα τα νέα μέλη και όσοι, όσοι δεν θέλουν να μην έρθουν. Θέλω λοιπόν να σε ευχαριστήσω και γι' αυτό επιπλέον γιατί πάντα θέλησες να αντιμετωπίσεις αυτούς οι οποίοι θέλανε προνομιακή αντιμετώπιση, κάτι το οποίο δεν άρεσε πολύ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα πράγματα έχουν αλλάξει φυσικά και θα ήταν καλύτερα να είχαν γίνει διαφορετικά. Τώρα, αν μιλήσουμε σε επίπεδο απολογισμού, βλέπουμε ότι οι τράπεζες χαϊδεύτηκαν ουσιαστικά και αντιμετωπιστήκαν με μεγάλη επίοικια μέσα στην κρίση και το κοινωνικό στοιχείο ουσιαστικά παραμελήθηκε. Πιστεύω ότι αν ήσουν πρόεδρος της Κομισιόν θα είχε αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα και θα είχε αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη ενεργητικότητα. Κάτι ακόμα το οποίο λείπει είναι και η συμμετοχή των πολιτών. <clears throat> και τώρα είναι παράξενο να <clears throat> το λέω έτσι. Πιστεύω ότι θα είχες προχωρήσει πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να, δώσει δυνατό, να μπορεί να δοθεί δυνατότητα στον πολίτη της Ευρώπης να θεωρήσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι το δικό του εγχείρημα. Και πραγματικά το ερώτημα είναι γιατί δεν είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα Juncker στην κεφαλή της. Σου εύχομαι λοιπόν όχι μονάχα να έχεις μια μακρά ζωή και ευτυχισμένη ζωή, αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο, να εξακολουθήσεις να είσαι ενεργός και ελπίζω ότι θα υπάρξει πάντα η ευκαιρία το 2014 να είσαι ο νέος πρόεδρος της Κομισιόν. Ίσως δεν είμαι τόσο ε, <laughs> αντικειμενικός όπως ο Σφεν Γίγκολτ, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ρωτώ αν συμφωνείς με αυτά ή όχι. Ναι. <laughs> Να προσθέσω και το εξή, λέει ο Ζαν ότι η συζήτηση έχει το αντικειμενικό της κομμάτι Εγώ χαίρομαι για όλους τους επένους. Νομίζω ότι έχουμε τους λόγους για τους οποίους έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει. Οι Γερμανοί πάντα θέλουν να γίνεται αυτό το οποίο είναι εφικτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι απαραίτητο να είναι κανείς πρόεδρος της Κομισιόν ή πρόεδρος του Συμβουλίου για να μπορέσει να, μπορέσει να ε, πείσει την Ευρώπη να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει πρέπει και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στις χώρες τους να υποστηρίζουν την Ευρώπη και όχι μονάχα όταν είναι στις Βρυξέλλες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η ευρωπαϊκή πολιτική δεν είναι ο Μπαρόσο, η Φανρομπά. Η ευρωπαϊκή πολιτική είναι καταρχήν αυτό που γίνεται μέσα στα εθνικά κράτη, μέσα στα εθνικά κοινοβούλια, μέσα στα κόμματα. η Ευρώπη πολλές φορές δεν είναι μέσα στα θέματα που συζητούνται σε εθνικό επίπεδο, αλλά αυτό πρέπει να γίνει. προσπαθώ να πάρω λίγο επιπλέον χρόνο από τους ε, διερμηνείς, ε, αλλά οι τρεις τελευταίοι, η Ντανούτα, η Σοφία και άλλος ένας, ε, κινδυνεύουν να μείνουν απ' έξω. Μάρκους Φέμπερ από το ΕΛΚ, παρακαλώ πολύ σύντομα. Και εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Το αντικειμενικό κομμάτι θα το συντομεύσω. Σα ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την εργασία σα. Δεν χρησιμοποιούμε όλη την ίδια παρτιτούρα στη Γερμανία θυμάμαι τις συζητήσεις που κάναμε το 2003-2004 σε σχέση με την ε, απάλυνση του πλαισίου σταθερότητας τότε και το αν όλα τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζονται με το ίδιο τρόπο και έρχομαι τώρα στο ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω. Λένε όλοι αυτό που είπες και εσύ ότι έχουμε ξεπεράσει το χειρότερο και εγώ συμφωνώ με αυτό. Παραμένει όμως το ερώτημα. Έχουμε διορθώσει όλα αυτά τα οποία έπρεπε να έχουμε κάνει ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη πρόκληση που μπορεί να προκύψει ή αν έχουμε ακόμα αντιμετωπίσει τα πιο σοβαρά αλλά δεν έχουμε ακόμα συμπληρώσει αυτό το πλαίσιο. Μήπως έχουμε ακόμα τον κίνδυνο με, την επόμενη, ε, με τον επόμενο κλειδονισμό είτε λόγω δημογραφικής αλλαγής είτε λόγω κάποιου άλλου λόγου να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Έχουμε χρησιμοποιήσει το καιρό της κρίσης για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα ή όχι. Αυτά τα οποία είπαμε τότε το 2003-2004 δεν αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό. Αυτά τα ξέρει και η Τσεσού και η Τσεντεού. Εάν είχαμε εφαρμόσει πλήρω το δημοσιονομικό πλαίσιο τότε, το πλαίσιο σταθερότητα, θα έπρεπε να είχαν υπάρξει και κυρώσει εναντίον τη Γερμανία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει τηρήσει κατά γράμμα το σύμφωνο σταθερότητας ήταν το Λουξεμβούργο. Ούτε και, ούτε και οι κατοχώρες Και οι κατοχώρες δύο φορές είχαν ξεπεράσει το όριο του, του πλαισίου του ελλείμματος. Μόνο το Λουξεμβούργο είχε τήρηση πλήρω το σύμφωνο σταθερότητα. Αλλά ξέρετε και το κάνει σαφές πάντα το κοινοβούλιο αυτό ότι έχουμε μια μεγάλη ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τα θέματα ρύθμισης στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ Δεν το έχει κάνει ούτε η Ευρώπη, δεν το έχει κάνει ούτε σε διεθνέ επίπεδο της κοινότητα και γι' αυτό είναι απαραίτητο να επισημαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι παραμένει ένα έλλειμμα στον τομέα αυτό. Εγώ είμαι πιο ήρεμος από ότι πέρσι, αλλά δεν είμαι ακόμα απόλυτα καθυσυχασμένος. Νομίζω θα ήταν καλύτερο για τον Γερμανό φορολογούμενο αν το 2003-2004 να είχαν εφαρμοστεί κάποια μέτρα και όχι τώρα να πρέπει να χρηματοδοτεί άλλες χώρες. Ναι, είναι πιθανό, λέει ο, ο Κατανοώ την απόψη αυτή. Ωραία, Άστριντ, Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα μια μικρή παρατήρηση όσον αφορά την πολιτική των ευκαιριών. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γιούγκερ. Δεν τον εκπλήσει αυτή η ευκαιρία που χάθηκε από την Επιτροπή μετά από 8 χρόνια προεδρία στο Eurogroup να μην υπάρχει μια γυναίκα επικεφαλής στην Ευρώπη. Άλλη ερώτηση τώρα. Γνωρίζουμε ότι η πολιτική λιτότητας δεν βοηθάει, οι άνθρωποι υποφέρουν τόσα εκατομμύρια συμπολίτε μας. Οπότε ποια πολιτική μείωση του ελλείμματος θα μπορούσαμε να έχουμε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το ότι υποφέρει ο κόσμος, οι πολιτικές αυτές έχουν οδηγήσει σε κάποια αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για πλήρη αποτυχία. Δεύτερον, είπατε στην εισαγωγή σας ότι για σας η κοινωνική διάσταση στην οικονομική και νομισματική μας πολιτική πρέπει να έχει σαν αποτέλεσμα ένα ελάχιστο επίπεδο κοινωνικών δικαιωμάτων ε, των ε, πολιτών μας. Ένα ελάχιστο μισθό για παράδειγμα. Ξέρουμε ότι ήταν 5% στον Οκτώβριο, ε, το 1η Ιανουαρίου άλλαξε τώρα. για να φτάσουν στα 1.024,19 για έναν ανεδίκευτο εργάτη και 1240 κάτι για έναν ε, εργαζόμενο με προσόντα, είναι ο ελάχιστος Αν έχετε έναν ελάχιστο κοινωνικό μισθό, αν υπήρχε δηλαδή αυτό στην Ευρωζώνη, ο πρόεδρος της Ευρωζώνης θα έπρεπε ίσως να κάνει κάποια παρατήρηση στην κυβέρνηση του Λουξεμβούργου για να υπάρχει κάποια συνοχή. Η αρχή ενό ελάχιστου κοινωνικού μισθού σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι κάτι που το θέλουν και άλλοι. Εγώ θα έπρεπε βασικά να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου που φρόντισε οι συνέπειες μερικές φορές καταστροφικές της κρίσης δεν έφτασαν στους ε, πιο δύναμους της κοινωνίας μας. Εντάξει, Άστριντ, δεν ξέρω αν είναι πραγματικά δικιά σου η παρατήρηση, αλλά δεν πρέπει να νομίζουμε ότι θα ήταν ε, καλό, σωστό και δίκαιο μια πολιτική λιτότητας που να απαιτεί τις μεγαλύτερες προσπάθειες από τους πιο αδύναμους. Εγώ θα ήθελα στην Ευρώπη τα βάρη, τις συνέπειες της κρίσης να τα επομισθούν οι πιο ισχυροί. Αυτό θα πει αλληλεγγύη μεταξύ ε, πολιτών σε μια κοινωνία. Όχι επειδή είναι περισσότεροι ή πιο αδύναμοι από τους πιο δυνατούς να επομίζονται εκείνοι τις συνέπειες μιας κρίσης. Εγώ βέβαια δεν στρέφομαι εδώ πέρα προς ε, έναν ε, ανόητο αριστερισμό, τέλος πάντων για να το πω έτσι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν δέχομαι μια τέτοια λογική. Δεν τη δέχομαι διότι πηγαίνει ε, προς ένα μοντέλο που δεν της Εγώ θέλω αλληλεγγύη. Θέλω οι πιο αδύναμοι να κάνουν και αυτή η προσπάθεια, αλλά αυτοί που δεν έχουν προβλήματα, που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα και που πλέον στον πλούτο, αυτοί επίσης να συνεισφέρουν στην συνολική προσπάθεια. Κατά τα άλλα, από το 1985 που είχαμε το σχέδιο Ντελόρ για την εσωτερική αγορά, εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το ελάχιστο κοινωνικό δικαίωμα. Έχουμε καταργήσει περίπου όλα τα εμπορικά εμπόδια. Έχουμε την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, πλήρως. Είναι απίστευτο στα κοινωνικά ζητήματα να έχουμε αγνοήσει μια προσαρμογή. Κάτι το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα σήμερα όλες οι προσπάθειες προσαρμογής που γίνονται, οι σχεδόν όλες, στοχεύουν το κοινωνικό επίπεδο. Είναι μια πολύ κακή αρχιτεκτονική αυτή που έχουμε στη βάση. Και αυτό το λέω τώρα, αλλά το έλεγα εδώ και 20 χρόνια. Και το λέω συνέχεια. Σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής ε, πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μήπως να μπορέσω να προτείνω το εξής, ε, να ομαδοποιήσετε τις ερωτήσεις και να απαντήσει μετά ο πρόεδρος Γιούγκερ, ε, γιατί είναι κρίμα. Είτε μερικοί δεν θα βάλουν τις ερωτήσεις τους, άλλοι ή δεν θα απαντήσει ο πρόεδρος. Πολύ ωραία. Ε, θα πάρουμε δύο ομάδες των τριών, έτσι. Πολύ ωραία. Θα δούμε αν θα λειτουργήσει καλύτερα. Ούντε Μπούρμαν. Θάρμαν. Και και μετά Ντανούτα, Άννη και Σοφή. Να δούμε αν μπορέσουν όλοι να μιλήσουν. Ούντο. Κύριε Πρόεδρε, θυμάμαι τα αρχικά σας λόγια που εκφράσατε την ε, ικανοποίησή σας γιατί το 2012 παρά τις προβλέψεις που είχαν γίνει δεν οδήγησε στη διάλυση της Ευρωζώνης. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό όταν βλέπουμε εκ των υστέρων τι έγινε. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μπει σε μια νέα κατάσταση <clears throat> όπου τα μελλοντικά προγράμματα βοήθειας δεν θα είναι ότι θα μπαίνετε το καλό είναι μάλλον ότι θα έχουμε ε, προγράμματα υποστήριξης τα οποία δεν θα λένε θα πάρετε χρήματα αν μειώσετε τον ελάχιστο μισθό, αλλά όταν θα έχετε προγράμματα τα οποία θα λένε καταπολεμήστε την φοροδιαφυγή, φτιάξτε καλύτερες δομές κτλ. Έχει λοιπόν αλλάξει η προγραμματική αντιμετώπιση των προγραμμάτων αυτών και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει αλλάξει την αντιμετώπιση τους. Όλα αυτά μας οδηγούν σε μια νέα μέθοδο εργασίας και ένα νέο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά με μια κοινή ε, αντιμετώπιση. Πώς θα βλέπατε να έχουμε μια κατάσταση όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συμφωνούν ότι τα εργαλεία, τα προγράμματα προσαρμογής, τα προγράμματα βοήθειας να έρχονται για συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής μας αυτή στον Ευρωπαϊκό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ζητούν και μία πλειοψηφία από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Αυτό θα ε, μας οδηγούσε να φύγουμε από αυτή την κατάσταση που οι αποφάσεις λαμβάνονται όλο και περισσότερο σε διακρατικό επίπεδο χωρίς ουσιαστικά τα εθνικά κοινοβούλια να μπορέσουν να ελέγξουν για τα θέματα αυτά. Δεν υπάρχει πια κοινοβουλευτικός έλεγχος έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Ο Διόγκο <coughs> τρέχει το ρολόι. Προσπαθήσουμε να είμαστε μέσα σε έξι λεφτά όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Σιάρον, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω κι εγώ <clears throat> με τα συγχαρητήριά μου για την εργασία σας ως επικεφαλής του, της Ευρωομάδας και να σας πω ότι είναι μια πραγματική ευγνωμοσύνη που νιώθουμε για σας και σας ευχόμαστε και μια μακρά πολιτική ζωή και από τη στιγμή που θα αποχωρήσετε από την Ευρωομάδα, από την Προεδρία του σε μια απάντηση που δώσατε στην Ελίζα Φερέιρα είπατε ότι τα κράτη τα οποία τηρούν τα υπεσχημένα στα προγράμματα σταθεροποίησης θα πρέπει να την χάνουν κάποια ανταμοιβή. Πώς θα μπορούσαμε να συγκεκριμενοποιήσουμε το θέμα αυτό. Αυτό έχει συζητηθεί ιδιαίτερα στην πορτογαλική κοινή γνώμη. Πώς θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η ανταμοιβή, μια επαναδιαπραγμάτευση των προγραμμάτων σταθεροποίησης, μια τροποποίηση αυτών των προγραμμάτων ή και ένα σύστημα το οποίο προβλέπεται να υπάρχουν ε, κίνητρα για τα κράτη αυτά που βρίσκονται σε μνημόνια για να τηρήσουν αυτές τις υποχρεώσεις που προβλέπονται. Θα ήθελα λοιπόν να έχω την απόψη σας. Ευχαριστώ όλοι. Κύριε Πρόεδρε, προετοιμάσατε ε, την, ε, τη διαδικασία της, ε, του ενιανομίσματος. Θα έχουμε και την Τραπεζική Ένωση, αλλά όπως είπατε και εσείς ο ίδιος, υπάρχουν και κάποιες φωνές που δεν είναι αρκετά βροντερές στην Ευρώπη και αναφερθήκατε στην έλλειψη κοινωνικού συμφώνου. Υπάρχει όμως μία μικρή φωνή στην οποία δεν αναφερθήκατε. Είναι ο προπολογισμό της Ευρωζώνης. Σε αυτό το κοινοβούλιο έχουμε ελάχιστες πληροφορίες, ε, αυτές που διαρρέουν στον τύπο μόνο. Και σας θέτω το ερώτημα, πού βρίσκεται η συζήτηση στο ε, Eurogroup. Τώρα που φεύγετε μπορείτε να μιλήσετε πιο καθαρά ίσως. Ε, ίσως μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω. Ξέροντας ότι σήμερα βλέπουμε ότι έχει εγγραφεί πλέον ε, η δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά δεν υπάρχει προπολογισμό τη Ευρωζώνης έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα ε, ασύμετρα σοκ και οι κρίσεις αυτέ. Με αισθάνομαι θυγμένος, αγαπητέ κύριε γιατί στην ουσία υπονοήσατε ότι μέχρι τώρα ε, χρησιμοποιούσα την ξύλινη γλώσσα των πολιτικών. Τώρα θα δείτε όμως τι σημαίνει ξύλινη γλώσσα. Εγώ είμαι υπέρ της εφαρμογής ενός αλληλέγγυου μηχανισμού ε, και εργαλείου στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Διότι υπάρχουν κάποιες κρίσεις, κάποια σοκ, τα οποία είτε έχουμε διανύσει ήδη, είτε προβλέπουμε να υπάρξουν που θα δημιουργήσουν ε, δημοσιονομικά προβλήματα, προβλήματα στον προπολογισμό ε, ενός ή περισσότερων κρατών μελών. Καλό λοιπόν ε, είναι να υπάρχει πέρα από τους μηχανισμούς FSF και ESM να, υπάρχουν, να υπάρχει και κάποιος άλλος μηχανισμός απορρόφησης των κραδασμών που προέρχονται από τέτοιου είδους κρίσεις ήταν μια πρόταση του Συμβουλίου αυτών των σοφών που αναφέραμε προηγουμένως, ε, την οποία όμως ε, δεν θεώρησε ορθή ε, και, το, και δεν συμπεριέλαβε στις προτάσεις το Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει όμως, τουλάχιστον όσον αφορά την ίδια την ορολογία, ε, έχουμε ε, αναφερθεί στο εργαλείο αλληλεγγύης που κατά την άποψή μου είναι ένας ε, σημαντικός δημοσιονομικός πυλώνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρωζώνη, δηλαδή και για τις χώρες μη Ευρωζώνης, έστω και αν είναι δύσκολο να επιτευχθεί η συμφωνία όλων αυτών. Αγαπητέ φίλε Φέιο, δεν μπορώ να σου πω εγώ ποιες θα είναι οι ανταμοιβέ ας πούμε που θα λάβουν ε, οι χώρες ε, οι οποίες οι αντισταθμίσεις, ε, οι χώρες οι οποίες θα έχουν προχωρήσει στα προγράμματα προσαρμογής με τρόπο πολύ ισχυρό όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία. αλλά αυτό που θέλω είναι να μην δώσουμε την εντύπωση ότι η Ευρώπη είναι μόνο τιμωρός. Η Ευρώπη είναι και αυτή η οποία θα ε, δείξει κατευθύνσεις, ε, η οποία ε, θα ανταμείψει προσπάθειες. Και για τον Ούντο ήθελα να πω το εξής, ότι δεν ισχύει ότι ζητήσαμε να εφαρμοστεί μονάχα μία πολιτική λιτότητος στα εργασιακά θέματα στις χώρες του Μνημονίου. Στην περίπτωση της Ελλάδος, εμείς πιέσαμε ιδιαίτερα να υπάρξει φορολογική δικαιοσύνη και να λειτουργήσει σωστά το φορολογικό σύστημα να γίνουν προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό λοιπόν θα γίνει και η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να χρησιμοποιήσει την βοήθεια της, ε, της Ευρώπης για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά το φορολογικό σύστημα. Και εγώ πράγματι <coughs> πιστεύω ότι δεν πρέπει απλώς να κηρύττουμε τη λιτότητα, αλλά να ζητούμε και υπευθυνότητα από τις χώρες που είναι αποδέκτρες των προγραμμάτων αυτών σταθερότητα. Το δεύτερο τμήμα τη ερωτήσεω θα το απαντήσω γιατί δεν με αφήνει η Πρόεδρος. Λυπάμαι, αλλά έχουμε πέντε λεφτά στη διάθεσή μα και έχουμε τρει ομιλητέ και πρέπει να αποχαιρετήσουμε και όλα τον Πρόεδρο. Ένα λεπτό ο καθένας σας. Δανιούτα, Ατι και Σόφη. Ευχαριστώ πολύ. Σαν Κλόντ, θα μου λείψεις και εμένα. Σου εύχομαι ότι το καλύτερο θα υπάρξουν προβλήματα. Και μια από τις κορυφές της κρίσης μπορεί να είναι μικρές τράπεζες. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, πώς θα αποφύγουμε μια τέτοια κατάσταση όπου μικρές τράπεζες να μην έχουν ε, υγιείς μηχανισμούς που να δίνουν εγγύησεις. Πώς θα το αποφύγουμε αυτό, αν υπάρξει πρόβλημα σε μια τράπεζα, ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό, δεύτερο σχόλιο. Θέλω να μας πεις ναι, ένα ισχυρό ναι. Για την κοινοτική μέθοδο στην Ευρωζώνη χρειαζόμαστε αλλαγή στη συνθήκη. Κατά τη διάρκεια της Λεξοβουργικής Προεδρίας είσαι διατεθειμένος να μας δώσεις μια νέα συνθήκη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ε, προσωπικά και εξ ονόματος των Ελλήνων πολιτών να σας ευχαριστήσουμε για τα όσα κάνατε για τη διαχείριση της κρίσης αλλά και κυρίως γιατί πάντα αντιταχθήκατε στις ε, στερεότυπες, ε, προκλητικές, υποτιμητικές πράξεις και δηλώσεις. Είστε πρόεδρος του Eurogroup από το 2005 και επομένως οι γνώσεις σας και οι εμπειρίες σας είναι πολύ βαθιές, όχι μόνο όσον αφορά την διαχείριση αλλά και όσον αφορά τα αίτια της κρίσης. Αν σήμερα σας ζητήσουμε πολύ σύντομα να καθορίσετε ε, τι θα μπορούσε να είχε γίνει με διαφορετικό τρόπο έτσι ώστε τα αρνητικά, οι αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης ε, να είχαν αποφευχθεί και όσον αφορά την πρόληψη και όσον αφορά τη διαχείριση. Τι θα μπορούσατε να μας πείτε. Ευχαριστώ πολύ. Σοφή, ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Γιούγκερ. Δύο ερωτήσεις έχω σύντομες. Είπατε ότι για να συμβουλέψετε το διάδοχό σας. Αγαπάτε τους άλλους και να τους ε, αντιμετωπίζετε σωστά. Αν δεν αγαπάει αλλήλους, τι θα γίνει τότε με την οικονομική μας ολοκλήρωση. Αν δεν επικυρωθούν αυτά που πρέπει να επικυρωθούν και αν δεν θέλει να ολοκληρώσει την Τραπεζική Ένωση. Αυτό θεωρείτε ότι θα ήταν αδυναμία του διαδόχου σας. Έπειτα λέτε ότι δεν θέλετε ένα τείχος ανάμεσα στις χώρες Ευρωζώνη και στις χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Πολύ συχνά όμως ξεχνάμε ότι εκτός από τις δύο εξαιρέσεις υπάρχουν και οχτώ χώρες οι οποίες έχουν δεσμευτεί ότι θα μπουν στην Ευρωζώνη. Τι γίνεται τώρα, έχουμε δεχτεί ότι δεν θα το κάνουν ποτέ ή γίνεται κάτι για να επιταχυνθεί η προσχώρησή τους στην Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ωραία, δύο λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Τυχερός είσαστε. Ευχαριστώ για την γενοδορία σας αυτή, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω στην Τανούτα ότι συμμερίζομαι τις ανησυχίες της. Δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι η συζήτηση που γίνεται και για τις αρχαί... την αρχή αυτή που λέει ότι πολύ μικρή, άρα δεν χρειάζεται βοήθεια. Αυτό είναι κάτι που όντως μας προβληματίζει και πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε για αυτό το σημείο. Θα έλεγα στην Ελληνίδα φίλη μας πως ναι. Ναι, όντως σε σχέση με την Ελλάδα και το ελληνικό έθνος πρέπει να σας πω ότι εγώ πάντα ένιωθα μια συμπάθεια και μια φιλία την οποία δεν συμμεριζόντουσαν πάντα οι φιλόσοφοι του Βορρά. Για μένα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη θα ήταν ατελείς χωρίς την Ελλάδα. Έχουμε γίνει αλαζόνες, δεν γνωρίζουμε την ιστορία και επειδή ακριβώς δεν αγαπάμε αυτούς που είναι και από μας, έχουμε την τάση να αγνοούμε αυτά τα οποία έχει προσφέρει η ελληνική δημοκρατία στην Ευρώπη και όσα έχουν προσφέρει οι Έλληνες. Εγώ θα στηρίζω αυτή την χώρα δεν θα έλεγα μέχρι το τέλος των ημερών μου, γιατί δεν θα είναι πάρα πολύ ίσως αυτό, αλλά αν μη τι άλλο να ξέρετε ότι είμαι φίλος των Ελλήνων και θέλω να είμαι φίλος όλων εκείνων που έχουν λιγότερους φίλους από τους μεγάλους. Και συνεχίζω. Μου ζητάτε να πω πράγματα, κυρία μου, για κάποιον που μπορεί να είναι ο διάδοχός μου, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι. Όποιος και να είναι λοιπόν, το ίδιο θα έλεγα. Στα 8 χρόνια που ήμουν επικεφαλής της Ευρωζώνης και μετά τα 30 χρόνια που ήμουν υπουργό, πολύ συχνά άλλαξα άποψη. Συχνά γιατί παρατηρούσα τους άλλους, προσπαθούσα να καταλάβω τους άλλους, προσπαθούσα να καταλάβω γιατί οι άλλοι λένε κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν περίμενα και τελικά πήρα μαθήματα ζωής. Αυτή είναι η πολιτική. Αν κοιτάτε μόνο τον εαυτό σας, αν ομφαλοσκοπείτε, αν είσαστε επικεντρωμένοι στη δικιά σας την καριέρα και φοβόσαστε να πείτε τα πράγματα όπως έχουν, χάνεται τελικά το νόημα της Ευρώπης. Στις χώρες μας έχουμε πει ότι πρέπει να υποστηρίζουμε την Ευρώπη και στην Ευρώπη πρέπει να υπερασπιζόμαστε τις χώρες μας. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Ο φιλόσοφος Πασκάλ είπε ότι εμένα μου αρέσουν τα πράγματα που πάνε μαζί, που συνδυάζονται καλά. Στην ε, Ευρώπη κινδυνεύουμε να χάσουμε τον μπούσουλα, αν δεν το κάνουμε αυτό. Πρόεδρο, Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά μας λείβει το ότι αποχωρείτε, γιατί πάντα χαιρόμασταν πάρα πολύ τις συναντήσεις μας. Περνάμε πάντα πολύ καλά. Τώρα εκ μέρους της Επιτροπής μας ολόκληρης θέλω να σας δώσω ένα μικρό δωράκι. Να, για να δούνε και όλοι τι είναι. Πρόκειται για ένα μετάλλιο, φαίνεται εδώ το ημικύκλιο, για να θυμόσαστε τι σημαίνει να έρχεται κανείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας το θορίζω λοιπόν και σας λέω κι εγώ πως θλίβομαι που αποχωρείτε. J'avais compris. Εγώ είχα καταλάβει ότι δεν χρειάζεται κανείς να είναι στο Eurogroup για να προσκαλείτε εδώ, οπότε θα ήθελα να σας ζητήσω να με προσκαλείτε κάθε μήνα. <laughs>